<laughs> Ladies and gentlemen, dear colleagues, let us begin. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε. Πρώτο θέμα για τη συνεδρίασή μα το απόγευμα είναι η ανταλλαγή απόψεων με τη Λετωνική Προεδρία Καλωσορίζω τον Υπουργό κύριο Ράσνα στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Θα συνεχίσω στα λετωνικά. Είναι τιμή η παρουσία μου σήμερα για να συμμεριστώ τις πρόοδες που επέτυχε η Λετωνική Προεδρία στο τομέα της δικαιοσύνης. Στην αρχή, όταν σας ενημέρωσα για τις δραστηριότητες του εξαμήνου μας, σας είπα ότι οι δραστηριότητες στην δικαιοσύνη συνδέονται όλο και πιο πολύ με την οικονομική ανάπτυξη, την ανάπτυξη, την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. Τη ενιαία εσωτερική αγορά. Γι' αυτό μια προτεραιότητά μας και καθήκον ήταν να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής Ευρώπης. λαμβάνοντα υπόψη αυτή την προτεραιότητα συνεχίσαμε την εργασία μας ακριβώς στον τομέα της δικαιοσύνης. Θέλουμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και να μειώσουμε την γραφειοκρατία είναι εξαιρετικά ουσιώδες να μειωθεί το κόστος των ενδίκων διαδικασιών, να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε τις ε, διασυνοριακές ένδικες διαδικασίες. Δικαιοσύνη για την ανάπτυξη λοιπόν είναι προτεραιότητά μας. Και ιδιαίτερα εστιάσαμε σε μια σειρά από προτάσεις να αναφερθώ σε ορισμένες. Τροποποίηση του κανονισμού για τη διαδικασία πτώχευσης. Μεταρρύθμιση για τα σήματα. Κανονισμός για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των δημοσίων εγγράφων. Τροποποίηση του κανονισμού για την επίλυση των μικροδιαφορών. Επίσης, σύσταση του Συμβουλίου για τη χρήση των βίντεο διασκέψεων. Επίσης τα δικαιώματα των μετόχων, η οδηγία γι' αυτό και οι μονοπρόσωπες εταιρείες. Και τέλος, θέματα που σχετίζονται γενικά με την μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα και πρόσβαση των τρίτων χωρών στη Σύμβαση της Χαΐς για τις ε, αστικές πλευρές των ε, απαγωγών παιδιών με μπλοκή διαφόρων χωρών. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μας γιατί επιτύχαμε αρκετά. Έρχομαι εδώ απευθείας από την ε, τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών στο Λουξεμβούργο και οι προγνώμονές μας πραγματικά έκαναν ό,τι μπορούσαν ούτω ώστε να προωθήσουμε όσο ήταν δυνατό διάφορα θέματα. Να ξεκινήσω αναφέροντας ότι μια βασική ημερομηνία ήταν η 13η Μαρτίου γιατί τότε το Συμβούλιο ενέκρινε την πολιτική συμφωνία με το Κοινοβούλιο για την τροποποίηση του κανονισμού για τη διαδικασία αφαιρεγγιότητας. Έτσι έχουμε ένα σύγχρονο μέσο για τις διαμεθοριακές διαδικασίες αφαιρεγγιότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ ότι ο κανονισμός αυτός θα δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στις ε, επιχειρήσεις που έχουν ε, προβλήματα ε, ταμιακά ούτως ώστε να αποφύγουν την πτώχευση και ε, να υπάρξει επίλυση των προβλημάτων τους. Στις 23 και 24 Απριλίου οργανώσαμε μία διεθνή συζήτηση για τον κανονισμό αφαιρεγγιότητας πρόσφατες τάσεις και προοπτικές. Διάφοροι πανεπιστημιακοί Ευρωπαίοι νομοθέτες και εκπρόσωποι κυβερνήσεων και ασχολούμενοι με τον κλάδο, επαγγελματίε του κλάδου δηλαδή, συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή και υπήρξε ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και προσεγγίσεων στις διάφορες χώρες, στον τομέα λοιπόν της αφαιρεγγιότητας. Ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι μαζί με εσά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταφέραμε να μεταρρυθμίσουμε τον τομέα των σημάτων. Το πακέτο για τα σήματα θα διασφαλίσει τον εξυγχρονισμό του συστήματος. Η καταχώρηση σημάτων θα είναι πιο προσβάσιμη για τις επιχειρήσεις το σύστημα γενικά θα γίνει πιο αποτελεσματικό και θα μειωθεί και το κόστος του. Σε σχέση με αυτό, ευχαριστώ ιδιαίτερα την κυρία Βίξτρα, δεν είναι παρούσα, αλλά την ευχαριστώ και ελπίζω να ενημερωθεί όταν θα ενημερωθεί για τις συνεδρίες. Για την προστασία των ε, διανοητικών δικαιωμάτων θελήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και 3 και 4 Μαρτίου οργανώσαμε μια συνδιάσκεψη για να αποκτήσουμε καλύτερη ενημέρωση για τις τάσεις για το θέμα αυτό στην ε, Λετωνία, την Ευρώπη, παγκοσμίω. Υπήρχε ευρεία αθρώα προσέλευση με ιδιαίτερα δικαιωμένους ε, καλεσμένους όπως ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Επίσης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σημάτων. Ήταν πραγματικά πολύ υψηλού επίπεδου η συμμετοχή. Μετά από μακροσκελής και περίπλοκες συζητήσεις μεταξύ των εμπειρογνωμόνων, χθες το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία για τον κανονισμό για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των εγγράφων. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένας συγκεκριμένος, πρακτικός τρόπος που θα διευκολύνει την κινητικότητα των εργαζομένων στην Ευρώπη και θα μας επιτρέψει να έχουμε έγγραφα για αστικά θέματα ευρωπαϊκά χωρίς επιπλέον γραφειοκρατία. Άρα η Ευρώπη θα γίνει πιο φιλική προς τους πολίτες της. Ελπίζω πολύ σύντομα να ξεκινήσει η διαδικασία τρεμερούς διαλόγου επ' αυτού και ότι στο εγγύς μέλλον θα είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε έγκριση αυτού του μέσου. Περαιτέρω. Διεξάγονται ακόμη τεχνικές και πολιτικές συζητήσεις για να βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ των, δικών σας, των σας ετοιμάτων και των ετοιμάτων του Συμβουλίου για την τροπολόγηση τη διαδικασίας επίλυσης μικροδιαφορών. Ελπίζω πράγματι να καταλήξουμε σε συμβασμούς κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες της Προεδρίας μας. Ως υπουργό Δικαιοσύνης θα αποτελούσε για μένα μεγάλη τιμή θα ήταν πραγματικά κολοφόν της Προεδρίας μας μια συμφωνία για μια απλουστευμένη προσέγγιση για τις διαμεθοριακές αστικές διαδικασίες. Και ευχαριστώ την κυρία Γκέρινγκ Όντεμπορντ για αυτό, για την εργασία που έχει ήδη επιτελέσει για το θέμα αυτό. Και λήξε στη δικαιοσύνη, πρέπει να ενθαρρύνουμε την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας. Για παράδειγμα, για τις διαμεθοριακές ένδικες διαδικασίες, η χρήση βίντεο διασκέψεων επιταχύνει τις διαδικασίες και μειώνει το κόστος. Γι' αυτό <clears throat> με χαρά σας ανακοινώνω ότι ενέκρινε το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης ε, τεχνικές συστάσεις για τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και συγκεκριμένα τηλεδιασκέψεων, βίντεο διασκέψεων και πιστεύω ότι με ταχύρυθμο θα προχωρήσουμε σε αυτό το τομέα. Η Προεδρία μας γνωρίζει παραδείγματα από διάφορες άλλες χώρες που αξιοποιούν τις ε, βίντεο διασκέψεις, όπως και στη Λετωνία τις χρησιμοποιούμε. Εάν τα δικαστήρια στην αρχή βέβαια ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικά, σήμερα ε, δεν υπάρχουν και τόσο πολλές επικρίσεις έναντι της χρήσης ε, αυτής της τεχνολογίας. Και αυτό έχει ήδη διευκολύνει την ε, πρόσβαση στη δικαιοσύνη και επίσης τη μείωση της καθυστέρησης εκδίκασης των υποθέσεων. Αυτό είναι λοιπόν ένα μέσο που μας βοηθάει και μας έχει βοηθήσει συγκεκριμένα στη Λετωνία σε αυτό το τομέα. Επίσης η Προεδρία μας ε, ε, ε έκανε μεγάλες προσπάθειες στο εμπορικό δίκαιο για να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό κλίμα και την ανταγωνιστικότητα. Στις 25 Μαρτίου θα κράτη-μέλη ενέκριναν τον συμβασμό της Λετωνικής Προεδρίας για, την οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων και αυτό μας επέτρεψε να εγκρίνουμε και εντολή για την έναρξη των τριμερών διαπραγματεύσεων. Ε, η διαδικασία αυτή επιτρέπει ευρύτερη συμμετοχή των μετόχων στη διοίκηση των ε, εισηγμένων εταιρεών. Κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία όπως είδαμε και κατά την πρόσφατη κρίση. Λαμβάνοντας υπόψη την σημασία του θέματος αυτού διοργανώσαμε στη Λετωνία μία διάσκεψη η εταιρική διακυβέρνηση και πώς θα προωθήσει την ανταγωνιστικότητα στην ψηφιακή εποχή. Και συζητήσαμε και τα προβλήματα που προανέφερα. Συζητήσαμε τις πρόσφατες εξελίξεις, τις τάσεις στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και άλλα θέματα που είναι σημαντικά για τους επενδυτές. Διοικητικά συμβούλια και επιτροπές ελέγχου. Το Συμβούλιο ανταγωνιστικότητα τη 28 Μαου, κατέληξε σε συμφωνία και ενέκρινε την εντολή για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις οδηγίες για τις μονοπρόσωπες εταιρείε. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που πιστεύουμε ότι θα διευκολύνει την ίδρυση εταιρεών και θα επιτρέψει την καταχώρηση των εταιρεών επιγραμμικά εταιριών με μετοχικό κεφάλαιο μόνο ενός ευρώ και ήταν προτεραιότητά μας να προωθήσουμε το θέμα αυτό. Φυσικά, για το θέμα αυτό, κάθε χώρα θα διατηρήσει κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες για να αποφευχθεί κατάχρηση αυτής της δυνατότητας. στη Λετωνία, ξέρετε. <clears throat> Έχουμε πολύ θετική εμπειρία μέσω της χρήσης αυτών των βελτιωμένων διαδικασιών και θα συνεχίσουμε να προωθούμε εξάλλου γενικά τη μεταρρύθμιση των δικαστηρίων για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών της Ένωσης προς τα δικαστήρια. Και το Συμβούλιο συμφώνησε στη διαδικασία για να διοριστούν επιπλέον δικαστές. Μόλις λοιπόν γίνει η μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Σας ευχαριστώ για όλη την ε, βοήθεια που μας δώσατε για το θέμα αυτό. Συνεργαστήκαμε καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου για να λάβουμε υπόψη τις απόψεις σας στα πλαίσια του τετραμερούς διαλόγου. Θέλαμε πάντα να καταλήγουμε σε κοινέ λύσεις. Στόχος μας ήταν πάντα να γίνονται συμφωνίες ε, ενωρίς για τη δεύτερη ανάγνωση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Δεν το επιτύχαμε πάντα, αλλά το Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να αξιοποιήσει αυτή τη δικασία στις 23 Ιουνίου στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης Υπουργών ε, Εσωτερικών Υποθέσεων. Ε, τώρα εφόσον μιλάμε για την ε, μεταρρύθμιση του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε το θέμα μακρόπνοα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δούμε προς τα πού θα εξελιχθεί δεν πρέπει να μας ε, περιορίζουν μόνο αυτά που θεωρούμε ότι θα συμβούν τα, τελευταία, επόμενα 4-5 χρόνια. Και πιστεύω ότι όσο ευρύτερα δούμε το θέμα αυτό, όσο πιο μάκρο πρόθεσμα, τόσο ταχύτερα θα καταλήξουμε στη συμφωνία ότι είναι αναγκαία αυτή η μεταρρύθμιση. Θα μπορούσε να υπάρξει και δικονομική μεταρρύθμιση βεβαίως, και μεταρρύθμιση όσον αφορά το προσωπικό του δικαστηρίου. Η Λετωνική Προεδρία μόλις χθε συμφώνησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει τη συμφωνία της Χάγης του 1998 για τις αστικές πλευρές της απαγωγής παιδιών της διασυνοριακής απαγωγής παιδιών στην ε, Ανδόρα και τη Σιγκαπούρη. Τα δικαιώματα των παιδιών είναι πολύ σημαντικά για μας και χαιρόμεθα που μπορέσαμε να προωθήσουμε την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στο διεθνές πλαίσιο. Τέλος, χθε είχαμε τη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο του Συμβουλίου μας. Ε, όλο αυτό το εξάμεινο ήταν για μένα και τιμή αλλά και πρόκληση. Και οδεύει τώρα προς τη λήξη της. Χαίρομαι για τα επιτεύγματα, φυσικά. Αλλά, αλλά, Λυπάμαι, λυπάμαι σε έναν βαθμό. Και έχω και ένα συνέστημα απογοήτευσης γιατί όλη αυτή η θαυμάσια ομάδα η οποία με πλαισίωσε και όλος αυτός ο όγκος εργασίας τον οποίο αντιμετωπίσαμε, όλη αυτή η πίεση θα χρειαστεί τώρα να αποτελέσουν παρελθόν. Αλλά θα έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την περίοδο της Προεδρίας μας και θα ευχόμουν πραγματικά ε, όλοι μας να είχαμε μια τέτοια εμπειρία. Είμαι πεπισμένος ότι η επερχόμενη Προεδρία του Λουξεμβούργου θα είναι τόσο αποτελεσματική και τόσο επιτυχημένη. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω τους κυρίους και, τις κυρίες και κύριους ευρωβουλευτές για τη συνεργασία, ευχαριστώ για την κατανόησή σας, για τις προτάσεις σας και για τη σημερινή τιμή που μου κάνετε με την παρουσία μου Ευχαριστώ πολύ. We thank Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για αυτή την ε, σαφή εικόνα των δραστηριοτήτων σας ε, στη διάρκεια του εξαμήνου. Πρόκειται βεβαίω για ανταλλαγή απόψεων, επομένως ε, θα ήθελα να ζητήσω από τα μέλη της Επιτροπής να παρέμβουν και να σχολιάσουν. Κυρία Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ ειλικρινά την Λετωνική Προεδρία Πρόκειται για μια πολύ αποτελεσματική και συγκεκριμένη προεδρία που εργάστηκε ιδιαίτερα αποδοτικά και θα ήθελα επίσης να τους ευχαριστήσω και για τον ενθουσιασμό τους, διότι ανέλαβαν τα καθήκοντά τους με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Για αυτούς ε, οι οποίοι θα αναλάβουν τα ενία θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα Ε, για όσους ε, δεν ήξεραν και τι να περιμένουν, ιδίω όταν πρόκειται για την πρώτη προεδρία, δεν έχουμε πολύ μεγάλες προσδοκίες στον τομέα αυτό. Ε, αλλά εγώ είχα την τύχη να συμμετέχω στον τριμερή διάλογο που αφορούσε ένα μεγάλο ε, πακέτο μέτρων, ένα θέμα το οποίο απασχόλησε και την Επιτροπή μας σήμερα το πρωί. Πρόκειται για ένα κανθόδε ζήτημα, πολύ δύσκολο. Ήταν ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε στη διάρκεια της Λετωνικής Προεδρίας. Ε, ευτυχώς ολοκληρώθηκε και αποτελεί πολύ μεγάλη ελπίδα για την επόμενη εβδομάδα ε, να περατωθούν οι συζητήσεις ε, την επόμενη εβδομάδα στον τριμερή διάλογο. Πρόκειται για τις μικροδιαφορές. Βέβαια δεν περιμένω και θαύματα από πλευρά σας, διότι ακόμα πόρα απέχουμε από την άποψη του Συμβουλίου. Η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαφέρει. Γνωρίζω βέβαια ότι έχετε ταλέντο στη διπλωματία και ελπίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι καλά. Να συγχαρώ και άλλη μια φορά λοιπόν την Προεδρία και χαίρομαι που είχα την τύχη να συνεργαστώ με μια τέτοια ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Mr. Karim. Ο κύριος Καρίμ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ που κάνατε τον κόπο να έρθετε εδώ στην Επιτροπή μας σήμερα και χαίρομαι ιδιαίτερα για το σημαντικό έργο και τις δράσεις ε, οι οποίες ανελήφθησαν από την ε, Λετωνική Προεδρία τους προηγούμενους μήνες. Υπάρχουν δύο ζητήματα επί των οποίων θα ήθελα κάποιες περαιτέρω πληροφορίες από πλευρά σας. Ελπίζω έτσι να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε και λίγο καλύτερα τι ακριβώς θα κάνουμε στο μέλλον. Το ένα αφορά ένα ζήτημα το οποίο ε, αυτή τη στιγμή είναι εξελίξη για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τον ε, διορισμό των δικαστών. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια ακριβώς θέση έχει το Συμβούλιο από αυτού και πού θεωρείτε εσείς ότι υπάρχει περιθώριο ε, ταχείας ευελιξίας. Ποιες ήταν ε, οι ελλείψεις ε, βάσει των συζητήσεων που θεωρειτε εσεις οτι υπαρχει περιθωριο ε ταχειας ευελιξιας ποιες ηταν οι ελλειψεις βασει των συζητησεων που καταφερε να κάνει η Προεδρία σας. Και δεύτερον, Σαφώς αυτή τη στιγμή υπάρχει χάσμα μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούμε να αναλάβουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα έχουν πολύ μεγαλύτερο λόγο στα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τις συζητήσεις όμως που έχετε κάνει εσείς στη διάρκεια της Προεδρίας σας Υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσατε να δώσετε εν είδη συμβουλής ε, για να ε, ξέρουμε πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε τα συγκεκριμένα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Είχα δει ε, παρουσίασή σας σε κάποια άλλη επιτροπή στην οποία ήμουν σκιώδης ε, εισηγητής και μπόρεσα να παρακολουθήσω και το έργο σας στη διάρκεια αυτού του εξαμήνου. Λυπάμαι που πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός. Πραγματικά. Ε, τα πάντα φάνηκαν να τρέχουν. Και εγώ συνεργάστηκα με την Προεδρία σας για ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα, αλλά πρόκειται για μια πολύ καλή ευκαιρία για να φανεί για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει κοινά ενδιαφέροντα για τις 28 χώρες. Υπάρχει αυτή η μοναδική ευκαιρία να συνεργαστούν οι χώρες μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά προκειμένου να αποφευθούν αυτές οι αποστάσεις μεταξύ πολιτών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αναφέρομαι ε, στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα για την ε, Συνεργασία και ελπίζω να ολοκληρωθούν την επόμενη εβδομάδα οι συζητήσει για τις επίλυση μικροδιαφορών, διότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο δεν επιλύθηκε ακόμα. Όλα όσα έχουν να κάνουν με θέματα εργατικού δικαίου. Παραδείγματο χάρη, ένας εργαζόμενος ο οποίος εργάζεται σε άλλο κράτος μέλος υπήκος άλλης χώρας μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί ε, να προσφύγει στη χώρα του ε, κατά του πρώην εργοδότη του. Υπάρχουν κάποιες ε, χώρες οι οποίες διαφωνούν με αυτή τη διαδικασία διότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι θα δεχτούν μια νέα μορφή σκλαβιάς. Κατά την άποψή μου, εγώ δεν θεωρώ ότι ένας Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να εργάζεται χωρίς να έχει στη συνέχεια το δικαίωμα να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του. Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά τα δικαιώματα. και 26 και 28 συγγνώμη χώρε μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα να προστατεύουν τους πολίτες τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας ενώνει ε, πέρα από τις δυσκολίες μας. Όπως έλεγε και η κυρία Γκέριγκερ, ε, αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν τα ενία της Προεδρίας μετά από εσά θα έχουν πάρα πολλή δουλειά. Σας ευχαριστώ. other... Δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητάει το λόγο. Ίσως ε, θέλετε να απαντήσετε κύριε Υπουργέ στις ερωτήσεις που σας ετέθησαν. Ναι, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, για τις ερωτήσεις. Καταρχάς, ευχαριστώ και πάλι κυρία Γκέριγκερ. Σας ευχαριστώ για την επικοδομητική συνεργασία μας και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αντίστοιχα παρά το γεγονός ότι θα αλλάξει ο δικός μου ρόλος, δεν θα είμαστε πλέον Προεδρία, αλλά ελπίζω να υπάρχει επικοδομητική συνεργασία και στο μέλλον ε, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Να περάσω στην ερώτηση του κυρίου ε, Καρίμ για τη γενικότερη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτημα, όπως θα γνωρίζετε βεβαίως. Αφενός, βραχυπρόθεσμα θα μπορούσε ίσως να θεωρήσει κανείς ότι πρέπει για ένα μέτρο το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και δεν θα αποφέρει καρπούς στο εγγύς μέλλον για την Ευρώπη, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι κοντόφθαλμη άποψη και θα πρέπει να το εξετάσουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το ζήτημα. Εάν ε, όντως το εξετάσουμε έτσι και με μακροπρόθεσμο όραμα, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι ο αριθμός των υποθέσεων και η καθυστέρηση των υποθέσεων έχουν αυξηθεί σημαντικά. Έχουν μειωθεί βέβαια πρόσφατα οι, ε, οι υποθέσεις, οι νέες υποθέσεις που υποβάλλονται, αλλά η καθυστέρηση των υποθέσεων που εκκρεμούν είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη. Και αυτό σημαίνει ότι και οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις πλήττονται και μπορεί ορισμένες φορές να έχουν και απώλειες ε, δισεκατομμυρίων ευρώ και ε, πολλές φορές οι απώλειες αυτές μπορούν να αντισταθμιστούν με όνο εάν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου. Γεγονός που σημαίνει ότι ουσιαστικά τους προσφέρουμε κάτι με το ένα χέρι και τους το στερούμε με το άλλο χέρι. Και αυτή είναι μια διαπανηρή διαδικασία. Ο τρόπος που διεξάγεται η διαδικασία αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα δαπανηρός, διότι καθυστερούν πάρα πολύ οι υποθέσεις και δεν μπορούμε να περιορίσουμε με ε, διαδικαστικές μεταρρυθμίσεις και μόνον. Θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των δικαστών. Ξέρω ότι ε, πολλές χώρες ισχυρίζονται ότι δεν είμαστε τόσο πλούσιοι ώστε να ε, ε, πληρώσουμε το τίμημα. Υπάρχει μια παροιμία στη χώρα μου που λέει ότι ο άπλιστος πληρώνει δύο φορές και νομίζω ότι αυτή εξηγεί πολύ καλά την κατάσταση. Χρειαζόμαστε ένα καλύτερο σύστημα. Εάν δεν προσαρμόσουμε το σύστημα μακροπρόθεσμα, η κατάσταση θα επιδενωθεί. Θεωρώ ότι αυτή είναι η μόνη λύση. Αρχικά 12 δικαστές ε, θα έχουμε πρώτα το αστικό δικαστήριο, μετά θα έχουμε το, το γενικό δικαστήριο και εκεί θα έχουμε 9 επιπλέον ε, δικαστές. Συνολικά θα έχουμε 28 δικαστές. Αυτό είναι το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα. Και επίσης τι θα γίνει με το προσωπικό του δικαστηρίου. Ε, αν θα υπάρξει αύξηση ή μείωση του προσωπικού, θα το δούμε μετά ε, τη μεταρρύθμιση. Αφού συμφωνηθεί η μεταρρύθμιση του δικαστηρίου, μπορεί να πρέπει να αυξηθεί και ο αριθμό των γλωσσομαθών νομικών ή κάποια άλλα τμήματα να μειώσουν το προσωπικό του. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αφήσουμε στου ίδιου του δικαστέ να το αποφασίσουν. Αυτά λοιπόν μπορώ να σα πω όσον αφορά τη μεταρρύθμιση αυτή. ο τετραμερής αυτός διάλογος που αναφέρα προηγουμένως δεν προχωρά τόσο καλά όσο περιμέναμε και ε, εξ όσου γνωρίζω το θέμα θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Υπουργών ε, Γενικών Υποθέσεων. Ε, αν δεν κάνω λάθος έχει προγραμματιστεί για κάποια από τις επόμενες συνεδριάσεις Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων αλλά ο, μέχρι τώρα ο τετραμερής διάλογος δεν ήταν τόσο ομαλός όσο περιμέναμε και θα πρέπει ίσως να βρούμε μια άλλη μορφή συνεργασίας και συζήτησης. Όσον αφορά τώρα το χάσμα μεταξύ πολιτών και θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, Το θέμα αυτό έχει σχέση και με τη νομοθετική μας διαδικασία, πόση διαφάνεια υπάρχει, πόσο επικαιροποιημένε οι διαδικασίες είναι, πόσο προβλέψιμε είναι και πόσο ενδιαφέρουν του ίδιου του πολίτε. Το ερώτημα είναι ε, κατά πόσον ε, οι πολίτες που παρακολουθούν ε, διαδικτυακά αυτή τη συνεδρίαση θα λάβουν απαντήσεις στις ερωτήσεις τους. Ίσως και ναι, αλλά πολλοί από τους Ευρωπαίους πολίτες δεν γνωρίζουν καν πώς ξεκινά η νομοθεσία, δεν γνωρίζουν τις διαδικασίες που διέπουν το νομοθετικό έργο πριν υπάρξει οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση και δεν γνωρίζουν αν οι πρωτοβουλίες οι οποίες ε, αποτελούν τη βάση της νομοθετικής διαδικασίας, είναι κάτι, το οποίο έχει ξεκινήσει τελείως αμερόληπτα ή έχει ξεκινήσει μετά από ε, πιέσεις από λόμπι. Υπάρχουν χώρες που δραστηριοποιούνται περισσότερο, παραδείγματος χάρη οι σκανδιναβικές χώρες είναι ιδιαίτερα δραστήριες, ζητούν περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη ενημέρωση από αυτών. Ε, κυρίως όσον αφορά τις νομοθετικές διαδικασίες και την προέλευσή τους. Ε, και πρέπει σίγουρα να γίνουν κάποια πράγματα από αυτόν. Η τελευταία ερώτηση είναι λίγο πιο περίπλοκη. Η ερώτηση του κυρίου Μπούντα για το δικαίωμα ε, των εργαζομένων. Υπήρχε και μία ερώτηση για τη διαδικασία επίλυσης των μικροδιαφορών και μετά έχουμε τα εργασιακά δικαιώματα. Η συζήτηση είναι εξελίξη με τα κράτη-μέλη για το θέμα της επίλυσης των μικροδιαφορών και δυστυχώς τα πράγματα δεν προχωρούν τόσο γρήγορα όσο θα περιμέναμε. Τα κράτη-μέλη πιστεύουν ότι υπάρχουν ανάγκες για μια πολύ σοβαρή αξιολόγηση των επιπτώσεων ε, για το ζήτημα αυτό. Ε, θα πρέπει να βρούμε ένα συμβιβασμό, αλλά προφανώς ε, αυτό το θέμα θα το προχωρήσει η Προεδρία του Λουξεμβούργου. Η πολύ καλή βοηθός μου λέει ότι ε, ελπίζουμε βέβαια να υπάρξει συμφωνία. Έχουμε ελάχιστε εβδομάδε μέχρι τι αρχέ Ιουλίου, αλλά ε, τίποτα δεν είναι απίθανο. Αυτά όσον αφορά τη διαδικασία επίλυση μικροδιαφορών. Τώρα, δικαιώματα εργαζομένων, νομίζω ότι λίγο πολύ τα κάλυψα αυτά. Δυστυχώ, κύριε Μπούντα, δεν ε, είμαι πλέον αρμόδιο για να θίξω το συγκεκριμένο θέμα σήμερα. αναφέρθηκα λίγο σε κάποια γενικά ζητήματα, ε, το πώς μπορούμε να μειώσουμε το χάσμα μεταξύ πολιτών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και αυτά από την πλευρά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Αυτό λοιπόν κύριε Υπουργέ, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω εσάς και τους συναδέλφους σας για όλη τη δουλειά που κάνατε το τελευταίο εξάμεινο σχεδόν. Πιστεύω πως η Επιτροπή μας εκτιμά το έργο που κάνατε εσείς και οι συναδελφοί σας ως κάτι πάρα πολύ θετικό και έχετε την ευγνωμοσύνη μας λοιπόν για αυτήν την καλή συνεργασία και είμαι σίγουρος ότι ακόμα και μετά την Προεδρία σας η συνεργασία μας θα εξακολουθούσε να είναι εξαιρετική. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για όλα όσα έχετε κάνει.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 Uh, Αγαπητά μέλη, η κυρία Γκένιγκερ διατύπωσε ένα αίτημα. Αν συμφωνείτε κι εσείς, θα εξετάσουμε τώρα το σημείο 30 της ημερήσιας διάταξης, Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών, γιατί η κυρία Γκέρινγκεν έχει ανεγκλημένε υποχρεώσεις αργότερα. Είμαστε λοιπόν στο σημείο 30 της ημερήσιας διάταξης και κυρία Γκέρνια έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση, συνόψιση του τελευταίου τρεμερού διαλόγου που έγινε πρόσφατα, ενώ ο επόμενος θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη. Και ελπίζουμε λοιπόν και αν ελπίζουμε είναι γιατί και η Λετωνική Προεδρία μας στηρίζει στην προσπάθεια που κάνουμε και στην ελπίδα που έχουμε να κλείσουμε μέχρι την ερχόμενη Τρίτη το θέμα αυτό. Πολλά θέματα έχουν ήδη ρυθμιστεί με τρόπο που μας ε, ικανοποιεί. Οπότε δεν θα τα πω όλα, δεν θα αναφερθώ σε όλες τις λεπτομέρειες. Απλώς θα αναφέρω το τεχνικό τμήμα, γιατί το πολιτικό τμήμα ούτως ή άλλως θα πρέπει να εκδεθεί σε πολιτικό επίπεδο. Πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσω ότι υπάρχει προφανής βούληση συνεργασίας από πλευράς του Συμβουλίου και η Λετωνική Προεδρία όντως έχει ασκήσει πιέσεις επί των κρατών μελών. Έκανε πολλά, ούτω ώστε να υπάρξει τάχιστα συμφωνία. Αύριο θα έχουμε μια άτυπη συνάντηση όπου θα μάθω ποιε είναι οι πραγματικές δυνατότητες που έχουμε να γίνουν αποδεχθέ οι θέσει μας από το Συμβούλιο. Αλλά όπω σα είπα, όλα θα εξαρτηθούν από τον τελευταίο τριμερή διάλογο, που ελπίζω λοιπόν να είναι ο τελευταίος, για την ερχόμενη Τρίτη. Τώρα, για τη διαδικασία. Είναι μια νέα διαδικασία που θα είναι στη διάθεση των ε, πολιτών. Και το καινότομο είναι, το, η καινοτομία συγγνώμη, είναι ότι προβλέπουμε ένα όριο πολύ ψηλότερο. Προηγουμένως ήταν 2.000 ευρώ. Τώρα το ανεβάσαμε στις 10.000 ευρώ, ούτω ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή τη νέα δυνατότητα στις διαφορές που έχουν ιδιαίτερα τις διαμεθοριακές. Αυτό το νέο όριο λοιπόν 10.000 ευρώ δεν αρέσει το Συμβούλιο και κατά πάσα πιθανότητα το Συμβούλιο δεν θα αποδεχθεί αυτό το νέο όριο άρα η εναλλακτική μας είναι 5.000 5.000 για τους ε, καταναλωτές, τα μονομένα άτομα και 5 με 10.000 για τις επιχειρήσεις. Ίσως να συμφωνήσουμε μόνο για το όριο των 5.000 και μεταγενέστερα να καταφέρουμε να το αυξήσουμε. Αλλά φυσικά δεν έχουμε ακόμη χάσει κάθε ελπίδα ότι θα αποδεχθεί το Συμβούλιο και τα δύο αυτά νότατα όρια. Αυτό θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τις βιντεοδιασκέψεις τώρα. Ο κύριος Υπουργός το ανέφερε και εκείνος το θέμα αυτό. Πολλά δικαστήρια τώρα σε πολλά κράτη-μέλη έχουν ήδη τον αναγκαίο εξοπλισμό για να ε, λαμβάνουν χώρα αυτές οι βίντεο διασκέψεις. Πρέπει λοιπόν να αφήσουμε ένα περιθώριο για την προσαρμογή, για τον εξοπλισμό σε όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον θα απαιτούμε να υπάρχει δυνατότητα χρήσης αυτών των νέων τεχνολογιών. Όμως το Συμβούλιο μέχρι στιγμής ε, δεν έχει ε, εκφράσει άποψη για τις συγκεκριμένες προθεσμίες. Πόσα χρόνια δηλαδή θέλουν για τον εξοπλισμό των δικαστηρίων. Θέλουμε εμείς να καθοριστούν σαφώς αυτά τα χρονικά όρια, αυτές οι προθεσμίες. Γιατί αν δεν ορίσουμε προθεσμίες, τότε ίσως αυτές οι νέες τεχνολογίες να μην ε, εγκατασταθούν ποτέ στα δικαστήρια, οπότε το θέμα αυτό ποτέ δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Ένα άλλο θέμα το οποίο ανέφερε τώρα και ο καθηγητής ε, Μπούντα. Αναφέρθηκε σε ορισμένα θέματα εργασιακού δικαίου. Θα θέλαμε αυτή η απλουστευμένη διαδικασία επίλυσης μικροδιαφορών να μπορέσει να συμπεριλάβει και σε ένα μικρό βαθμό το εργατικό δίκαιο. Για παράδειγμα, αν ένας εργαζόμενος ε, δεν έχει πληρωθεί, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτή η διαδικασία έναντι του ε, εργοδότη. Επειδή βεβαίω ο εργαζόμενο είναι αδύναμος έναντι του, ε, ο εργαζόμενος είναι αδύναμος έναντι του εργοδότη, θα θέλαμε λοιπόν να έχει πρόσβαση σε αυτή την απλούστερη διαδικασία. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε όλοι σας τη διαδικασία σε όλες τις λεπτομέρειες. Θέλουμε αυτή η διαδικασία να είναι απλή, απλουστευμένη, να μην απαιτεί να μετακινηθεί κάποιος για να παραστεί ενώπιον ενός δικαστηρίου, ούτω ώστε να μειωθούν και τα δικαστικά έξοδα, γενικότερα το κόστος δικαιοσύνης και να επιτρέπει την επίλυση των μικροδιαφορών, γιατί αλλιώς ε, διαπιστώνουμε ότι οι μικροδιαφορές ε, τελικά ε, δεν αξίζει τον κόπο για κάποιον να απαιτήσει να επιληθούν γιατί το κόστος της επίλυσης ε, υπερβαίνει το όφελος, ε, το αναμενόμενο όφελος, την αναμενόμενη αποζημίωση, αμοιβή κτλ. που δεν έχει λάβει ακόμη. Για τα έξοδα της δικαιοσύνης γενικότερα και τα δικαστικά έξοδα συγκεκριμένα. Είπαμε ότι θα πρέπει να μην υπερβαίνει το 5% του ύψους του ε, υπο ε, εξέταση ποσού, υπο, υπο απαιτούμενου ποσού, συγγνώμη αλλά ε, ορισμένα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν. Δεν θα θέλαμε όμως ε, το θέμα αυτό να είναι μόνο αρμοδιότητα των κρατών μελών. Θα θέλαμε να υπάρξει μια αναλογική σχέση μεταξύ των δικαστικών εξόδων και του απαιτητού ποσού. Γιατί τι έννοια θα έχει για παράδειγμα τα δικαστικά έξοδα να είναι 50% του ποσού το οποίο διεκδικεί κάποιος. Τότε φυσικά κανείς δεν πρόκειται να μπει σε αυτές τις περιπέτειες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα λογικό ποσοστό μεταξύ του απαιτητού ποσού και, το, και των δικαστικών εξόδων. Να είναι ένα ποσοστό δηλαδή το ένα το άλλο. Και κάτι τελευταίο που ήθελα να υποβάλω είναι το θέμα της κατεξοδότησης πράξεων. Εμείς, ε, μάλλον να το πω αλλιώς, προβλέπεται η δυνατότητα των κατεξοδών της πράξεων γιατί αυτό επιτρέπει βεβαίως δυνατότητες αυτόνομης δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά μόνο για τεχνικές προσαρμογές. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε κάτι τέτοιο. Οι κατοξιδότητες πράξης είναι ίσως οι πιο κατάλληλες για τις τεχνικές ε, προσαρμογές των κειμένων. Κατά την πρώτη μας συνάντηση με το Συμβούλιο, το Συμβούλιο αρνήθηκε συνολικά την δυνατότητα κατά εξοδότηση πράξεων. Ήθελε μόνο εφαρμοστικές. Τώρα η κατάσταση έχει κάπως αλλάξει και νομίζω ότι γίνονται πιο αποδεκτές οι κατεξοδότες συμπράξεις και ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα να καταλήξουμε να επικυρώσουμε σε αυτή μας την προσέγγιση που ήταν η αρχική μας προσέγγιση. Και κάτι τελευταίο, θέλαμε να εφαρμόσουμε το πεδίο εφαρμογή αυτής της δυνατότητας σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις δυσφήμισης. Δηλαδή, στις περιπτώσεις δυσφήμισης, ξέρετε ότι πολύ συχνά οι αποζημιώσεις ε, που απαιτούνται ε, ξεπερνούν τις 5-10.000 ευρώ. Γι' αυτό σκεφτήκαμε να υπάρχει μια ταχύη διαδικασία για περιπτώσεις δυσφήμισης ε, στο διαδίκτυο, για παράδειγμα, να κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ των ε, πιο ελαφρών ας πούμε, και βαρύτερων περιπτώσεων. Όμω το Συμβούλιο δεν συμφωνεί γιατί οι διαδικασίε είναι πολύ διαφορετικέ από κράτο μέλο κράτο μέλο και αυτή η δυνατότητα να επεκτείνουμε τη ε, διαδικασία αυτή και για τη δυσφήμιση θα πρέπει να καταληφθεί η προσπάθειά μα αυτή γιατί το Συμβούλιο δεν θα το δεχτεί ποτέ. Καλύτερα να προσφέρουμε μια δυνατότητα που να μπορεί να αξιοποιηθεί από τους καταναλωτές, από τις μικρομεσαίες, παρά να είμαστε πιο αισιόδοξοι και τελικά να μην αλλάξουμε την κατάσταση τη σημερινή που δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Γενικά πιστεύω ότι έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας προτείνω λοιπόν να δεχθούμε αυτή τη δυνατότητα. Δεν είναι τέλεια, αλλά θα υποχρεώναμε την Κομισιόν να κάνει σε μερικά χρόνια επίσης μία εξέταση να δει αν μπορεί να αυξήσει τα όρια και να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σε ενημερώσω πριν από τον επόμενο λοιπόν τριμερή διάλογο που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη και ευελπιστώ ότι τα περισσότερα αιτήματά μας, ε, επιδιώξεις μας θα γίνουν δεκτά από το Συμβούλιο και την Λετωνική Προεδρία, η οποία μας είπε ότι και εκείνη ελπίζει ότι θα είναι δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε κάποιος να πάρει το λόγο. Μάλιστα. Εξαγγλίσατε το θέμα. Επομένως, νομίζω πως τελειώσαμε με αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γκέρνιερ. Έχω και ένα παρόμοιο αίτημα από τον κύριο Καρίν, ο οποίος θα ήθελε το δικό του σημείο εξέταση τροπολογιών σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα να συζητηθεί τώρα και μου υποσχέθηκε πως θα είναι πάρα πολύ σύντομος, αν κατάλαβα καλά. και οι εκλέκτοι καλεσμένοι μας συμφώνησαν. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Κύριε Καρύμ, έχετε το λόγο. Να είμαι υπόχρεος και σε εσάς, κύριε Πρόεδρε και στους προσκεκλημένους για τη χάρη αυτή που μου κάνετε. Δεν θα μακρηγορήσω καθόλου, φυσικά. Το θέμα αυτό συζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που κατέβαλαν κόπο και χρόνο για να συνεισφέρουν στο σχέδιο έκθεσης. Πολλές τροπολογίες πιστεύω θα ενισχύσουν την έκθεση και είναι μάλιστα αποτέλεσμα ενός διαλόγου που λαμβάνει χώρα και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε διαφορετική άποψη και διαφωνούμε, όμως ωστόσο πιστεύω να μπορέσουμε να βρούμε κάποιον κοινό τόπο μία λύση είτε σήμερα είτε στην ε, συνάντηση των σκιωδών εισηγητών που έχω προτείνει να γίνει πάρα πολύ σύντομα. Κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρετε, πιστεύω πως η επικουρικότητα και η αναλογικότητα πρέπει να θεωρούνται αναπόσπαστο στοιχείο, αφετηρία αν θέλετε, οποιασδήποτε πολιτικής. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε εάν οι στόχοι πολιτικής θα ε, πραγματοποιηθούν καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλές φορές η δράση σε παγκόσμιο επίπεδο είναι προτιμητέα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν απαιτείται καθόλου κάποια δράση. Δεν θα επαναλάβω τώρα εδώ όλα τα σημεία που ανέφερα στη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών, όμως θα ήθελα να τονίσω ορισμένα σημεία. Καταρχάς δεν πιστεύω πως ε, πρέπει να φοβόμαστε την έννοια της επικουρικότητας, διότι η επικουρικότητα μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε το δημοκρατικό έλλειμμα και να συμπεριληφθούν τα εθνικά κοινοβούλια ε, από την αρχή μιας διαδικασίας. Φυσικά έχουμε επίγνωση των διάφορων προβλημάτων εφαρμογής στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε από την αρχή να συμπεριλάβουμε τα εθνικά κοινοβούλια έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στο ε, αρχικό του στάδιο, παρά να έρθουμε αντιμέτωποι με ένα διεγκωμένο πρόβλημα αργότερα. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, ενδιαφέρουσες προτάσεις από τους συναδέλφους σε διάφορες ε, προηγούμενες συζητήσεις και εδώ στην Επιτροπή και ζητήθηκε να καλέσουμε διάφορους εθνικούς εμπειρογνώμονες ή να διοργανώσουμε βιντεοδιασκέψεις έτσι ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή τους, όπως προβλέπεται άλλωστε από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έχει προταθεί ένας μόνιμος εισηγητής από αυτήν την Επιτροπή. Και στην ε, πρότασή μου προτείνω μία διαδικασία κόκκινης κάρτας έτσι ώστε τα Εθνικά Κοινοβούλια να είναι σε θέση να εκφράσουν τις ε, ε, σκέψεις τους ή τις αμφιβολίες τους ε, για την αναλογικότητα ή για διαδικασία σε και οι απαντήσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων θα πρέπει να είναι ε, δυνατόν να εξετάζονται έτσι ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία. Επίσης, προτείνω μια διαδικασία πράσινης κάρτας όπου τα Εθνικά Κοινοβούλια θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροπολογίες ή να ανακαλούν ευρωπαϊκή νομοθεσία. Από ό,τι βλέπω από τις τροπολογίες υπάρχει κάποιος δισταγμός ε, για τις προτάσεις αυτές και θα ήθελα να μάθω τους λόγους για αυτόν τον δισταγμό και γι' αυτό λοιπόν προτείνω κάποια ιδιαίτερη συνάντηση έτσι ώστε να καταφέρουμε να βρούμε ένα συμβιβασμό. Προσωπικά πιστεύω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη συμπερίληψη των εθνικών κοινοβουλίων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα μπορούν να ασκούν βέτο σε ευρωπαϊκά μέτρα. Πρέπει όμως να σεβόμαστε το δικό τους ρόλο και να στηριζόμαστε στην ε, συμμετοχή τους και στη στήριξη των ε, νομοθετικών ε, προτάσεων. Γι' αυτό λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα με μεγάλη μου χαρά να ακούσω τα σχόλιά σας, είτε σήμερα είτε αργότερα, και τις προτάσεις σας για το πώς μπορούμε να προωθήσουμε το έργο αυτό. Όπως σας είπα, σκοπεύω να διοργανώσω μια συνάντηση σχεδόν εισηγητών πριν την ψηφοφορία στην Επιτροπή, έτσι ώστε να ε, ανταπεξέλθω σε όλες τις ε, ερωτήσεις και απορίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελε κάποιος το λόγο. Κύριε Κάουφμαν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον εισηγητή μας Μα επέστησε λοιπόν την προσοχή σε αυτές τις ε, πολλές τροπολογίε που έχουν υποβληθεί, πολλές από αυτές από εμένα. Και θα ήθελα να αναφερθώ σήμερα σε ορισμένα από αυτά. Καταρχάς πρέπει να ομολογήσω ότι όταν διάβασα την έκθεση μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι ο εισηγητή έχει κάπως ε, επικριτική άποψη για την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ταυτόχρονα όμως μου δημιουργήθηκε και η εντύπωση ότι έχει μείνει προσκολλημένος στις συνθήκες, εξέταση της επικουρικότητας και μόνο σε αυτές. Και αυτό το κάνει σε αρκετά σημεία, τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται, σε σημείο μάλιστα που δεν προχωράει η έκθεση εξαιτία αυτού. Και θα σα αναφέρω ορισμένα παραδείγματα. Είδα τα νούμερα από το Γερμανικό Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, που αναφέρονται στην επικουρικότητα, στην εξέταση της επικουρικότητας από το Γερμανικό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια. Σε τέσσερα λοιπόν χρόνια, 440 μία νομοθετικές προτάσεις της ε, Κομισιόν ε, παραπέμφθηκαν στην Bundestag για εξέταση και 157 περιπτώσεις εντοπίστηκαν όπου χρειάστηκε λεπτομερής εξέταση. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι το Γερμανικό Κοινοβούλιο σε αυτά τα τέσσερα χρόνια Μόνο τρεις από αυτές τις 441 ε, περιπτώσεις ε, παρέπεμψε πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό λοιπόν μας δείχνει ότι η επικουρικότητα και η αναλογικότητα τηρούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους. Τώρα, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για τα Εθνικά Κοινοβούλια πιστεύω πως θα είναι αρκετά δύσκολο να ε, Και αυτές οι 8 εβδομάδες πραγματικά δεν φτάνουν, πιστεύω. Και ταυτόχρονα αυτό το παράδειγμα του Γερμανικού Κοινοβουλίου μας δείχνει ότι γίνεται να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα των 8 εβδομάδων. Επίσης, έχει συζητηθεί το ότι θα μπορούσαμε για την εξέταση της επικουρικότητας να χρησιμοποιήσουμε και άλλα μέσα να αναφέρω ενδεικτικά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει πράσινες και λευκές βίβλους, κάποιες γνωμοδοτήσεις από τα Εθνικά Κοινοβούλια, δημόσιες διαβουλεύσεις, ε, από τα Εθνικά Κοινοβούλια επίσης. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες να εξετάσουμε το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον. Με άλλα λόγια, τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν πολλές δυνατότητες μέσα σε αυτές τις 8 εβδομάδες να ε, ολοκληρώσουν το έργο τους. Επίσης, αν δούμε το σύνολο του έτους, στις εργασίες των ε, κοινοβουλίων, θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν πολλές μέρες τις οποίες δεν συνεδριάζουν τα κοινοβούλια και Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται κάποια ευέλικτη ερμηνεία αυτού του χρονοδιαγράμματος. Αυτό όμως που πιστεύω ότι δεν πρέπει να αλλάξει είναι οι προθεσμίες στις συνθήκες. Πιστεύω επίσης πως ε, θα μπορούσαν να ανακυψούν πολλά προβλήματα στην εσωτερική λειτουργία των Εθνικών Κοινοβουλίων κατά τη διάρκεια αυτή τη διαδικασία εξέταση, τη επικουρικότητα. Και αυτό γιατί διαφέρουν τα Εθνικά Κοινοβούλια από κράτο μέλο σε κράτο μέλο. Α δούμε για παράδειγμα την περίπτωση Αυστρία και Γαλλία. Οι Ευρωπα... Ε, Επιτροπές Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αναλαμβάνουν εκεί τις ε, εξετάσει επικουρικότητα. όμως το γερμανικό κοινοβούλιο, τις οι περιπτώσει αυτές εξετάζονται ε, ανάλογα με τον τομέα της κάθε επιτροπής. Έπειτα, η εισαγωγή μιας ε, διαδικασίας κόκκινης και πράσινη κάρτας. Εδώ πρέπει να πω ότι η πρόταση αυτή δεν με βρίσκει σύμφωνη και δεν μπορώ να τη στηρίξω. Τα εθνικά κοινοβούλια ελέγχουν τις κυβερνήσεις τους και πιστεύω πως οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν υποχρέωση ενώπιον των κοινοβουλίων τους να τους ενημερώνουν για τις εργασίες και για ό,τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Και πιστεύω πως το δικαίωμα πρωτοβουλίας συμπερασματικά χρειάζεται να παραμείνει δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό μεταξύ άλλων αναφέρομαι στις δικές μου προτάσεις και στο δικαίωμα ανάκλησης σε Είχαμε και μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με αυτό, το δικαίωμα πρωτοβουλίας και το δικαίωμα ανάκλησης των ε, νομοθετικών προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τέλος πιστεύω ότι αυτά που λένε οι συνθήκες σχετικά με την ε, διαδικασία και ο ρόλος που έχει το κάθε θεσμικό όργανο δεν πρέπει να αλλάξει αντιθέτως με, αντίθετα με αυτά που προτείνει ο εισηγητής και την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων. Πιστεύω πως πρέπει να παραμείνουμε και να διατηρήσουμε μάλλον τους ε, ρόλους των θεσμικών οργάνων έτσι όπως ε, προβλέπονται από τις ε, συνθήκες πριν προβούμε σε αλλαγή τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ ο κύριος Άντερσον. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να μιλήσω σου ειδικά. Ναι, ωραία. Εμένα μου αρέσει η πρόταση αυτή. Περιλαμβάνει πολλές καλές ιδέες και σίγουρα αξίζει τον κόπο να τις επεξεργαστούμε περαιτέρω. Ιδίω την πρόταση για μια πράσινη κάρτα. Θεωρώ ότι είναι πολύ επικοδομητικός τρόπος ε, να ε, ε, εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή πολιτική και να την προσεγγίζουμε στους πολίτες. Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες βελτίωσης. Με αυτή την πρόταση για την κόκκινη κάρτα, βάσει της οποίας ε, κάποια κοινοβούλια κρατών μελών μπορούν να σταματήσουν μια διαδικασία, δεν είμαι εξίσου ενθουσιώδης. τα πάντα βέβαια θα εξαρτηθούν και από τη διαδικασία που θα αποφασίσουμε να εγκρίνουμε. Μετά έχουμε την κίτρινη κάρτα, και εδώ νομίζω ότι προσφέρονται περισσότερες δυνατότητες για βελτιώσεις. Αυτή τη στιγμή ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν ε, χρησιμοποιείται η κίτρινη κάρτα είναι γιατί υπάρχει ένα όριο για να ξεκινήσει η χρήση της και είναι τόσο υψηλό το όριο που πολλά κοινοβούλια δεν ε, θα επενδύσουν ε, έργο, το έργο που απαιτείται ώστε να γίνει ο έλεγχος της επικουρικότητας. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να μειωθεί το όριο και το χρονοδιάγραμμα που έχει ένα κοινοβούλιο ώστε ε, να μπορέσει να κάνει τον έλεγχο να παραταθεί. Εάν μπορέσουμε λοιπόν να μειώσουμε το όριο ε, και αυξήσουμε το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και να μην χρειαστεί αλλαγή της συνθήκης. Θεωρώ ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα και θα μπορούσαμε ίσως να την εξετάσουμε λίγο περαιτέρω. Ε, υπάρχει και αυτή η ιδέα των αξιολογήσεων των επιπτώσεων. Δεν έχω κάτι εναντίον των αξιολογήσεων επιπτώσεων αυτών καθεαυτών, πρόκειται για κάτι καλό, αλλά πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην έχουμε υπερβολικά πράγματα. Εμεί είμαστε πράσινοι και οι πράσινοι ε, δρούν. Θέλουν το Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση και να βελτιώσει λίγο τα πράγματα. Γι' αυτό και μα ανησυχεί ε, το γεγονό ότι τελικώ μπορεί να έχουμε πολύ περισσότερε αξιολογήσει επιπτώσεων. Διότι οι αξιολογήσει επιπτώσεων εξετάζουν την ποιότητα και εάν ε, εξετάσουμε μόνο το κόστο για τι επιχειρήσει και δεν μπούμε στον κόπο να εξετάσουμε και ποια είναι τα πιθανά ωφέλη για την κοινωνία. Για παράδειγμα, εάν ε, υπάρξει κάποιος καθαρισμός που θα βελτιώσει το περιβάλλον. Τότε μπορεί να έχουμε ε, λιγότερη και φτωχότερη νομοθεσία, διότι τα πάντα θα ε, παρακολύονται από την υπερβολική γραφειοκρατία. Ε, δεν θα θέλαμε λοιπόν να εγκρίνουμε ελαφρά την καρδία ε, περισσότερες αξιολογήσεις επιπτώσεων καθήκον μα είναι να έχουμε καλή νομοθεσία και τώρα και στο μέλλον. Σε γενικές γραμμές όμως θεωρώ ότι η έκθεση είναι καλή και θέλω να προχωρήσει και να την επεξεργαστούμε περαιτέρω. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ε, έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποια σχόλια από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο έκθεση και τι τροπολογίε, διότι παρά το γεγονό ότι η έκθεση περιλαμβάνει αρκετέ καλέ ιδέε, περιλαμβάνει και κάποιε προβληματικέ προτάσει. Τέσσερι παρατηρήσει θα κάνω. Η πρώτη είναι μια διευκρίνηση. Όταν η έκθεση προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τη την αιτιολογημένη γνώμη που λαμβάνει από τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, ως δέσμη ε, ε, προτάσεων ως συνέχεια μιας αιτιολογημένης νόμης. Αυτό είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Ε, όσον αφορά τις συνέπειες για την επικουρικότητα, κάθε νομοθετική πρόταση που έχει υποβληθεί σε αιτιολογημένη γνώμη ε, καταγράφεται σε κατάλογο και από εκεί και πέρα κάθε αιτιολογημένη γνώμη ε, αντιστοιχείται με την αντίστοιχη νομοθετική πρόταση ακόμα και αν η αιτιολογημένη γνώμη εξετάζει μια δέσμη προτάσεων. Νομίζω ότι με αυτή τη διευκρίνηση ε, στην πραγματικότητα συμφωνούμε πλήρως με αυτό το οποίο ζητούν κάποιες τροπολογίες μία αιτιολογημένη γνώμη που εκφράζεται ως τμήμα, ε, ως ε, ένα σύνολο κάποιων προτάσεων, ε, λαμβάνεται υπόψη όπως και μία μεμονωμένη αιτιολογημένη γνώμη για μία πρόταση. Επίσης, έχουμε κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος της κίτρινης κάρτας που είναι ενισχύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19 Μαΐου υπέβαλε μια δέσμη μέτρων για την καλύτερη νομοθεσία, η οποία σημαίνει ότι οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσουν την ποιότητα των αιτιολογήσεων που δίνονται στα επεξηγηματικά σημειώματα κάθε νομοθετικής πρότασης, ακριβώς για να εξηγήσουν καλύτερα σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια και ε, περαιτέρω σε όλους τους ενδιαφερομένους πώς ανταποκρίνεται η πρόταση στην αρχή τη επικουρικότητα. Τώρα, ε, οι πιο προβληματικές συστάσεις. Καταρχάς, ε, η δημιουργία νέων ε, καρτών. Βέβαια, πάντα πρέπει να υπάρχουν νέε ιδέες, αλλά πρέπει να είμαστε και σαφεί. Κάποιε ιδέες για πράσινες ή κίτρινε κάρτε μάλλον πράσινε ή κόκκινε κάρτε, απαιτούν αλλαγή τη συνθήκη. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί από μόνη τη να ερμηνεύει το πρωτόκολλο 2 για την επικουρικότητα με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που αναφέρεται στη συνθήκη και επιβεβαιώνεται και από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και για την επέκταση της προθεσμίας των 8 εβδομάδων. Οι προθεσμίες δυστυχώς ε, καθορίζονται βάσει νόμου και είναι προθεσμίες που πρέπει να γίνονται σεβαστές. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερμηνεύει ευνοϊκά ή αρνητικά ε, προθεσμίες, ε, για παράδειγμα στον τομέα του ανταγωνισμού ή των κρατικών ενισχύσεων, κανείς δεν θα δείξει κατανόηση και νομίζω το ίδιο ισχύει και εδώ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση η συνθήκη λέει 8 εβδομάδες, αλλά θα σας δώσουμε 10 ή 12 εβδομάδες. Δεν γίνεται. Η ιδέα μιας πράσινης κάρτας ε, εξετάζεται αυτή τη στιγμή από τα Εθνικά Κοινοβούλια και τα ίδια τα κοινοβούλια αντιλήφθηκαν ότι ίσως να μην πρόκειται για τη σωστή έννοια. Η ιδέα είναι ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να συνομιλούν και να δουν ποιες προτεραιότητες θα πρέπει να αντανακλώνται στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις τελευταίες συζητήσεις στην Επιτροπή Κόζακ, που είναι ο φορέας ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα εθνικά κοινοβούλια, χρησιμοποιήθηκε η ορολογία να ενισχύσουν τον πολιτικό διάλογο που σημαίνει ότι θα μπορούν να προτείνουν ε, πράγματα τα οποία θα μπορούσε να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας της και αυτή είναι μια εξέλιξη της έννοιας της πράσινης κάρτας μεν, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνεται ε, πλήρως σεβαστό το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τελευταία παρατήρηση είναι μια πολύ ευαίσθητη, κάτι το οποίο προτείνεται στο σημείο 14 ε, της, ε, του σχεδίου έκθεσης. Πρόκειται για αυτή την περίοδο αναμονής ε, βάσει της οποίας ε, τα, στο τέλος μιας διαδικασίας βάσει της οποίας θα υπάρχει ένα διάστημα αναμονής μέχρι να γίνει η αξιολόγηση επιπτώσεων και κάποιος έλεγχος και σας ευχηθώ την προσοχή εδώ. Υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες, κυρίως ε, για τη δεύτερη ανάγνωση και τη διαδικασία συνδιαλλαγής, οι οποίες μπορεί να μην συνάδουν πλήρως με αυτές τις νέες ιδέες και το γεγονός ότι αυτές οι ιδέες είναι αρκετά αντιφατικές ε, ε, εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή έχουν μιλήσει οι συνομοθέτες στον τριμερή διάλογο, αυτό σηματοδοτεί και το τέλος της διαδικασίας και όχι την έναρξη μιας νέας διαδικασίας. Ενδιαφέρουσες λοιπόν οι ιδέες, αλλά θα πρέπει να τις εξετάσουμε και από πολιτικό και τεχνικό πρίσμα, διότι υπάρχουν προθεσμίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένε στη συνθήκη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σα ευχαριστώ, κύριε Δεν βλέπω να θέλει κανεί άλλο το λόγο. Ο κύριος Βιέσκα, ο σκιώδης του ΕΛΚΑ, μου ζήτησε να σας αναφέρω ότι ζητάει συγγνώμη που δεν μπορεί να παρευρεθεί και προσβλέπει στην συνεργασία με όλους τους ε, ενδιαφερόμενους. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να... Α, συγγνώμη πως ο κύριος Καΐν θέλει να αντιδράσει. Αν όχι, μπορούμε να κλείσουμε αυτό το θέμα. Ο κύριος Καρίν. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Για να πω κάτι για να διευκρινίσουμε δύο-τρία θέματα από τους συναδέλφους ε, που τέθηκαν τους συναδέλφους και από την Κομισιόν. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν τον λόγο και συνέβαλαν στη συζήτηση σήμερα. Είμαι σίγουρος ότι στις συναντήσεις με τους Κιώδης θα σημειώσουμε ουσιώδη πρόοδο για όλα αυτά τα θέματα που ετέθησαν. Κυρία Κάφμαν, Αναφερθήκατε στην εμπειρία του Γερμανικού Κοινοβουλίου, αλλά δεν είναι η ίδια η πείρα, φοβάμαι, σε άλλα κοινοβούλια. Και αυτό ήδη το έχω συζητήσει απευθείας με τα Εθνικά Κοινοβούλια, για να τα ενθαρρύνω να κυκλοφορήσουν οι βέλτιστες πρακτικές. Και το δικό σας κοινοβούλιο θα μπορούσε να παίξει ηγετικό ρόλο για να αξιοποιήσουμε αυτές τις πρακτικές και αλλού γιατί κάνει πολλά για να υπάρξουν βελτιώσεις που μου αρέσουν. Καταλαβαίνω αυτά που Κομισιόν για το θέμα των προθεσμιών. Το έθεσε και η κυρία Κάφμαν και άλλοι συνάδελφοι επίση. Και αυτό το συζήτησα απευθεία σε επαφέ με τα Εθνικά Κοινοβούλια και στις συναντήσεις με την κόζα και αλλού. Και εκφράστηκε σαφέστατα η άποψη ότι η αυστηρή εφαρμογή της προθεσμίας 8 εβδομάδων τους δένει τα χέρια σε διάφορες φάσεις διαδικασίας ανάλογα με το Κοινοβούλιο και ζήτησαν έντονα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τόσο ώστε σε αυτή την περίοδο να λαμβάνονται υπόψη οι κοινοβουλευτικές διακοπές, τα καλοκαίρια, θεομηνίες που μπορεί να συμβούν, που επηρεάζουν και την εργασία του Κοινοβουλίου και των κυβερνήσεων, αν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη με κάποιο τρόπο. Και στρεφόμενος προς την Κομισιόν, πρέπει να πω ότι με ενθαρρύνει πολύ η προσέγγιση του Αντιπροέδρου Τίμερμαντς, που ήρθε και με είδε πριν οριστεί Επίτροπος και συζητήσαμε αναλυτικά μια σειρά από αυτά τα θέματα και πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα με βάση το πρόγραμμα εργασιών που μας έχει αποσταλεί υπάρχει λοιπόν ουσιώδες πιθανότητα να προωθήσουμε μερικές από αυτές τις ιδέες με έναν πολύ καινοτόμο τρόπο και ορισμένα από αυτά που υπόθηκαν από την Κομισιόν τα καταλαβαίνω απόλυτα καταλαβαίνω γιατί τα λένε αυτά αλλά δεν νομίζω ότι όλα αυτά τα αιτήματα θα οδηγήσουν ε, τα διέξοδα τα οποία ορισμένοι φοβούνται. Νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο κινητικότητα, Επανέρχομαι τώρα στο σύστημα κίτρινη, πράσινη, κόκκινη κάρτα. Είναι προτάσει. Θα τι συζητήσουμε αναλυτικά στι συναντήσει των σκιωδών και ευρύτερα ούτω ώστε να κάνουμε μόνο αυτό που τεχνικά λειτουργεί είναι συμβατό με τις συνθήκες και προτάσεις λοιπόν θέλουμε να προωθήσουμε που θα βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας και όχι να χαλιναγωγήσουν, όχι να δέσουν τα χέρια στη διαδικασία. Είναι απόλυτα επικοδομητική η προσέγγιση μου. Δεν θέλω να προωθήσω καθόλου κάποιες εθνικιστικές απόψεις. Νομίζω ότι όλα τα τελευταία χρόνια αυτό που έχω κάνει το αποδεικνύει αυτό και θα συνεχίσω να εργάζομαι προς αυτή την κατεύθυνση. Θα κάνω ό,τι μπορώ, ούτω ώστε όλοι οι συνάδελφοι να θεωρήσουν ότι μπορούν να υποστηρίξουν το τελικό κείμενο της εκθεσής μας όπως διαμορφωθεί εδώ στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτος, ευχαριστώ. Κλείνουμε λοιπόν το σημείο 28 και να περάσουμε στο 27. Να καλωσορίσω τους συναδέλφους μας από την Υπηρεσία Μελετών του Κοινοβουλίου, την Υπηρεσία Τεκμηρίωσης. Και να δώσω το λόγο στον κύριο Νταν να ξεκινήσει αυτή την παρουσίαση. Ευχαριστώ. Να κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή για να πω ότι το EPRS, η Υπηρεσία Ερευνών και η Διεύθυνση για τις μελέτες επιπτώσεων συντονίζει την στήριξη στην έκθεσή σας. Ε, όπως ξέρετε δημιουργηθήκαμε μετά από πρόταση της κυρίας Νίμπλε, χαίρομαι που είναι παρούσα. Βεβαίως έχουμε αναπτυχθεί πολύ από το 2011 που δημιουργηθήκαμε και αυτόματα καλούμεθα να βοηθήσουμε τέτοιες εκθέσεις για να υποστηρίξουμε την πολιτική, την, συγγνώμη, την προσέγγιση των κύκλων πολιτικής, να δούμε τι ελλείψεις υπάρχουν. Ιδιαίτερα τώρα εδώ που συζητάμε την οδηγία InfoSoc του 2001, για να καταλάβουμε καλύτερα τι πρέπει να κάνει τώρα ο νομοθέτης, να βοηθήσουμε το Κοινοβούλιο για τη συζήτηση για τις νέες νομοθετικές προτάσεις όταν θα υποβληθούν αργότερα φέτος. Τι κάνουμε λοιπόν. Παραγγέλνουμε διάφορες μελέτες και με βάση αυτές θα ετοιμάσουμε μια μελέτη επιπτώσεων που ελπίζουμε να συμποβάλουμε τον Ιούλιο. Σήμερα αυτό που σας παρουσιάζουμε είναι μια έκθεση προόδια από διάφορους τομείς. Θα ακούσετε τέσσερις παρουσιάσεις Έχουμε ήδη κάνει κάποιες παρουσιάσεις ε, για τα πνευματικά δικαιώματα. Θα ακούσετε τώρα από την Άταλη Βάλενς και πάρα από την Αντία Ράντελ για την εσωτερική αγορά και από τον Μάρτιν Γένσεν για τη βιομηχανία και τις βιομηχανικές σχέσεις. Αυτά είχα να πω μόνο. Να περάσουμε το λόγο στους εμπειρογνώμονες. Είναι εντυπωσιακοί οι εμπειρογνώμονες υψηλού επίπεδου. Έχουμε συνολικά 15 εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με αυτό το θέμα και στηρίζουν την εργασία της Επιτροπής σας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ. Ε, πάρτε το λόγο με τη σειρά που προτιμάτε. Να ξεκινήσω. Αντρέα Ρέντα. Είμαι στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών Πολιτικής θα παρουσιάσω ορισμένα θέματα την μόνη έκθεση που είναι σχεδόν ε, τελειωτική γιατί είναι εκ των υστέρων αποτίμηση της οδηγίας για την κοινωνία της πληροφορίας, InfoSoc. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για την εξάντε ανάλυση που γίνεται. Αλλά βασιζόμαστε και σε προηγούμενη εργασία που γίνει για την αποτίμηση εκ των υστέρων. Για να δούμε αν λειτουργεί. Η όλη ιδέα μιας αποτίμησης εκ των υστέρων είναι όπως θα δείτε να δούμε αν οι αρχικοί στόχοι συγκεκριμένων νομοθετημάτων επετέφθησαν κατά την εφαρμογή. Αν επετέφθησαν με αποτελεσματικό τρόπο, αν ε, τα νομοθετήματα και διατάξεις ε, είναι συμβατά και μεταξύ τους και με άλλα νομοθετήματα, άλλα τμήματα του κοινοτικού κεκτημένου. Και αν ακόμη εξακολουθούν να είναι χρήσιμα. Εδώ ασχολούμεθα με τα διανοτικά δικαιώματα στην επιγραμμική εποχή. Αυτό είναι πολύ επίκαιρο θέμα γιατί η τεχνολογία αλλάζει πολύ γρήγορα γιατί πιέζει τους νομοθέτες ε, να νομοθετούν με τρόπο που να συμβαδίζει με την τεχνολογία. Γιατί ξεκίνησε αυτή η οδηγία InfoShock. Υπήρχε ανάγκη να ευθυγραμμιστεί η νομοθεσία με τις δύο συνθήκες που είχαν υπογραφεί το 1996 στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και επίσης γιατί ήταν τμήμα των συνθήκων που διεύρυναν και ενίσχυαν τον ορισμό και την εφαρμογή των διανοητικών δικαιωμάτων στην ε, εποχή του ίντερνετ και στις απειλές που υφίστατο το copyright. γιατί όπως ξέρετε υπάρχουν πολλές απειλές ε, λόγω των δυνατοτήτων αντιγραφής, peer-to-peer, peer to peer που διευρύνονταν, διότι αυτό το νέο περιβάλλον, ε, πλήρως ψηφιακό, πλήρως από τελικό χρήστη σε τελικό χρήστη, αξιοποιείται όλο και περισσότερο από τους χρήστες. Άλλος στόχος ήταν, είναι, ήταν να εναρμονίσουμε τα πολλά νομοθετήματα που υπήρχαν και ακόμη υπάρχουν σε πολλά κράτη-μέλη. Γιατί αυτός ο καταγερματισμός είχε να κάνει όχι μόνο με συγκεκριμένα θέματα, αλλά και με το βασικό ορισμό των δικαιωμάτων, δηλαδή πώς ε, εφαρμόζονται όλα αυτά. Γιατί θεωρούνται αυτά τα δικαιώματα και ο τρόπος εφαρμογής εμπόδιο στην ε, ενιαία αγορά. Και επειδή αλλάζει το περιβάλλον στο ίντερνετ, θέλαμε να υπάρξουν και διατάξεις για να έχουμε μια δίκαιη αμοιβή των ε, δημιουργών και ε, ερμηνευτών. Τι κάναμε λοιπόν τότε. Επιλέξαμε μια νομική βάση που ήταν η μόνη δυνατή βασιζόταν στην ε, ανάγκη προσέγγισης νομοθεσιών. Τελικά αυτός δεν ήταν ε, ο κύριος στόχος της οδηγίας. Το πρώτο συμπέρασμα αποτίμησης μπορώ να σας πω ότι η οδηγία αυτή τελικά προσπάθησε να ενισχύσει και να διευρύνει τα πνευματικά δικαιώματα στα πλαίσια των υπαρχουσών συνθήκων αλλά με βάση μια νομική βάση που κυρίως ασχολείται με την εναρμόνιση και προσέγγιση της νομοθεσίας. Οπότε υπάρχουν πολύ διευρυμένα δικαιώματα, αλλά εφαρμόζονται ε, ιδιαίτερα αδύναμα. Άρα η εναρμόνιση είναι πολύ μικρότερη από ό,τι αναμέναμε. Άρα έχουμε περιορισμένη εναρμόνιση ακόμη και μεταξύ των βασικών ορισμών των δικαιωμάτων. Έχουμε αποκλίνοντες. Τα δικαιώματα τελικά καθορίζονται εθνικά έχουν να κάνουν με την αρχή της εδαφικότητας. Ακόμα και οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που είναι βασικό τμήμα αυτής της νομοθεσίας εφαρμόζονται και ερμηνεύονται πολύ διαφορετικά από κράτος σε κράτος. Όλος αυτός ο συνεχιζόμενος κατακαιρματισμός οδήγησε το δικαστήριο σε πυροσβεστικό ρόλο να προσπαθήσει να ενθαρρύνει τη σύγκληση όσον αφορά την εφαρμογή και ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξαιρέσεις και περιορισμούς. Αλλά αυτό ήταν υπερβολικό για το δικαστήριο. Σε πολλές περιπτώσεις έπρεπε να καλύψει κενά σε ένα ιδιαίτερα σαθρό περιβάλλον και επανειλημμένα επικρίθηκε το δικαστήριο και κατηγορήθηκε ότι υπερβαίνει τις ε, αρμοδιότητές του. Δηλαδή ότι προσπαθεί να δημιουργήσει νόμο μέσω της νομολογίας. Λοιπόν, όπως είπαμε είναι πολύ ε, ευρέως ε, καθορισμένα τα δικαιώματα και εφαρμόζονται αδύναμα. Γιατί είναι τόσο πλατιά διατυπωμένα, γιατί θέλαμε να διασφαλίσουμε την προστασία των δικαιωμάτων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους. Θέλαμε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα. Αλλά η προσπάθεια να τα προστατεύσουμε, να τα εφαρμόσουμε, συγκρούστηκε με ορισμένες άλλες θεμελιώδεις αρχές. Μία από τις αρχές αυτές είναι αυτή που είχαμε στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και με την προστασία των δεδομένων, το δικαίωμα της ιδιωτικής σφαίρας, το δικαίωμα λειτουργίας επιχείρησης. Όλα αυτά σε κάποια φάση διαπιστώσαμε ότι συγκρούονται με πολύ ε, διευρυμένες προσπάθειες να εφαρμοστεί η προστασία των δικαιωμάτων. Προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε το e-pred και τα ασφαλιστικά μέτρα στο αστικό πλαίσιο δεν έχουν βοηθήσει να εφαρμοστούν τα δικαιώματα. Και τα μέτρα τεχνολογικής προστασίας που θεωρούσαμε ότι ήταν πολλά υποσχόμενα τελικά δεν αξιοποιήθηκαν τόσο πολύ. Τα κράτη-μέλη δηλαδή έχουν ακολουθήσει διαφορετικές προσεγγίσεις για να εφαρμόσουν τα δικαιώματα ορισμένε φορέ μέσω διοικητικού δικαίου, δηλαδή κανόνε διοντολογία για παράδειγμα. Αυτό είχε επιπτώσεις για τη συνολική προστασία ε, ε, και λειτουργία του συστήματο. Άλλα προβλήματα τα τεχνικά μέτρα οδήγησαν σε ε, κατακαιρματισμό της αγοράς και επίσης η χορήγηση αδειών ε, ανάδικαιοδοσία όλα αυτά προσπαθούν να επιτύχουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ αυτό που θέλουν να εφαρμόσουν διαφορετική πολιτική τιμών από αυτούς που τελικά βλάπτουν τους τελικούς χρήστες. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα για τον νόμο για τα διανοτικά δικαιώματα και σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή για τις προσπάθειες καταπολέμησης των μονοπωλίων όπως για παράδειγμα στην περίπτωση Amazon. Ο άλλος στόχος που επιδιώξαμε είναι ότι παρά το ότι ένας από τους βασικούς στόχους της οδηγίας Infosoc ήταν η σωστή αμοιβή για τους δημιουργούς και ερμηνευτές. Τελικά το κείμενο της οδηγίας δεν περιέχει συγκεκριμένα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλα νομοθετήματα στον τομέα αυτό προσπαθούν τουλάχιστον να επιτύχουν αυτή την ε, σωστή αμοιβή αλλά ακόμη και σήμερα η κατάσταση των δημιουργών ερμηνευτών πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω. Και συνολικά η δυνατότητα που έχουν να απαιτήσουν σωστή αμοιβή οι δημιουργοί ερμηνευτές αφήνεται στις δυνάμεις της αγοράς. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Έχουμε λάβει μια σειρά ερωτήσεις από το Κοινοβούλιο που αναφέρονται σε αυτά που είπα στην αρχή. Πόσο αποτελεσματικό είναι το πλαίσιο αυτή τη στιγμή για να επιτύχει τους στόχους του, τους διατυπωμένους οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με λογικό κόστος. Και υπάρχει συμβατότητα ή είναι συνεπές εσωτερικά το πλαίσιο πολιτικής ή κάποια μέτρα αντιφάσκουν με ορισμένα άλλα και η εξωτερική συμβατότητα. Αυτό το πλαίσιο μήπως συγκρούεται με άλλα νομοθετήματα, με θεμελιώδεις αρχές και πόσο παίζει ακόμη το ρόλο του αυτό το πλαίσιο. Οι τεχνικές εξελίξεις όπως βλέπουμε έχουν αλλάξει την κατάσταση. Δεν τα είχε προβλέψει όλα αυτή η οδηγία. Μπορούμε να πούμε σήμερα ότι είχε αλλάξει τόσο πολύ ο κόσμος που να χρειάζεται να αλλάξουν κάποιες ρήτρε. Έχω εδώ ένα τμήμα του πίνακα αποτίμησης εδώ βλέπετε ότι σε μια κλίμακα από 1 έως 5 δεν έχουμε βάλει και πολύ ψηλούς βαθμούς ε, στο υπάρχον πλαίσιο. Από τα τέσσερα λοιπόν αρχικά κριτήρια της πρώτης διαφάνειάς μου μπορούμε νομίζω να ισχυριστούμε ότι μόνο το πρώτο η συμμόρφωση με το διεθνές νόμο εν μέρη έχει χωρίς βέβαια να λέμε πως δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Οι άλλοι στόχοι θα λέγαμε ότι σαφώς δεν έχουν επιτευχθεί. Τώρα για την αποτελεσματικότητα, σχέση κόστους αποτελέσματος, δεν μπορούμε να το επιτύχουμε αφού δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα. Αλλά ακόμη και η ανάλυση του κόστους η σημερινή κατάσταση κατακαιρματισμού δημιουργεί τρομερά, τρομερό κόστος, ε, νομική ανασφάλεια και διάφορους φραγμούς που μειώνουν κατά πολύ τη λειτουργία του παρόντος συστήματος για την ε, συνέπεια εσωτερική και εξωτερική σε διάφορες περιπτώσεις υπάρχουν προβλήματα η οδηγία αυτή βεβαίως από μόνη της είναι σχετικά συνεπές νομοθέτημα αλλά τελικά διαπιστώσαμε ότι συγκρούεται σοβαρά με άλλα νομοθετήματα ε, επίσης σημαντικά και τελικά ακόμη και κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει νομοθεσία δικαιωμάτων που υπερβαίνουν αυτή την οδηγία διότι αυτή η οδηγία και ο τρόπος που έχει εφαρμοστεί έχουν δημιουργήσει προβλήματα για την προστασία των δεδομένων, των εταιρών δικτύου. Είναι ακόμη λοιπόν κατάλληλη επιπλέον η οδηγία αυτή. Ναι, εξακολουθεί να είναι κατάλληλη να παίζει ρόλο για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Ζούμε σε μια πραγματικότητα που αυτό που πριν από λίγο θεωρείται ότι μπορούσε να προστατευτεί με τεχνολογικά μέτρα. Είμαστε τώρα σε ένα περιβάλλον όπου έχουμε πολλές δυνατότητες να κάνουμε streaming, να κατεβάσουμε η αξιοποίηση κειμένων και στοιχείων, η πρόσβαση σε περιεχόμενο και διασυνοριακά όλα αυτά καλούν για μία εκβάθρον επανεξέταση του παρόντος συστήματος των δικαιωμάτων. Τώρα πώς θα γίνει δεν μπορώ να σας πω τώρα γιατί υπάρχουν άλλες τρεις παρουσιάσεις αλλά αυτή η εκ των υστέρων μελέτη αξιολόγησης θέτει μερικά σημεία που ε, είναι καλά για την εκ των προτέρων επόμενη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ε, πω ότι η παρουσίαση σας στήρικε σε 15 λεπτά και δεν μας μένει λοιπόν πολύ χρόνος για τις επόμενες τρεις παρουσιάσεις. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να είμαστε σύντομοι. Νάταλη Μωρένης από το Μιλίο. Θα σας παρουσιάσω ορισμένα ευρήματα, προκαταρκτικά ευρήματα από το Πανεπιστήμιο του Μάστρικ και τις νομικές πτυχές της πνευματικής ιδιοκτησίας. Εστιαζόμαστε στα ωφέλη τη ε, οδηγίας και στι ε, δυνατότητες μεταρρύθμισης του συστήματος πνευματικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητήθηκε λοιπόν και πριν το θέμα, οπότε θα είμαι σχετικά σύντομη. Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τα Πνευματικά Δικαιώματα αποτελείται από 10 οδηγίες που δημιουργήθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια και υπάρχουν και διάφορες επιτυχίες στα πνευματικά δικαιώματα. Όπως ξέρετε, εγκρίθηκαν οι οδηγίες αυτές με στόχο να μειωθούν τα εμπόδια στην παροχή υπηρεσιών δεν πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μειονεκτήματα αυτού του κατακαιρματισμού είναι ότι υπάρχουν κενά στην νομοθεσία και έχουν προκύψει και νέε προκλήσεις. Η ψηφιοποίηση, για παράδειγμα, η εφαρμογή και το πλαίσιο τα πνευματικά δικαιώματα, το οποίο δεν ε, μπορεί να συμπεριλάβει όλες τις ε, περιπτώσεις, για παράδειγμα διαδικτυακή μετάδοση. Εδώ, εν συντομία, βλέπετε τα κύρια δικαιώματα και το βαθμό αναρμόνησής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως βλέπετε, τα περισσότερα είναι μερικώς αναρμονισμένα. Έχουν εναρμονιστεί μερικώς, για, για παράδειγμα, για ορισμένες περιπτώσεις το δικαίωμα επανάληψης, αναμετάδοσης, επίσης έχει εφαρμοστεί μερικώς. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις και ορισμένοι εθελοντικοί περιορισμοί. Δηλαδή η εφαρμογή διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο της απεραιτέρω εναρμόνισης και τι θα γίνει με τα υφιστάμενα κενά. Και προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε τις θετικέ και αρνητικές επιπτώσεις. Τις θετικές φυσικά είναι η βελτίωση της εσωτερικής αγορά, ε, η καλύτερη ασφάλεια δικαίου, καλύτερη σαφήνεια, μετά οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς οι περισσότεροι από αυτούς θα επωφεληθούν από την ε, περαιτέρω εναρμόνιση και ενσωμάτωση. Και λιγότεροι θα επιδεινώσουν και λιγότεροι δεν θα επωφεληθούν. Τώρα, πώς μπορούμε να συνεχίσουμε. Υπάρχουν τέσσερις δυνατότητες, όπως βλέπετε και τα πιθανά, οι πιθανές εξελίξεις. Κωδικοποίηση, νούμερο ένα. Η κωδικοποίηση τι σημαίνει. Η συγκέντρωση όλων των πτυχών σε μία νομοθετική πράξη. Εδώ υπάρχει η δυνατότητα αποσαφήνισης, διόρθωσης λαθών και δεν θα χρειαστούν ουσιαστικές αλλαγές στην νομοθεσία. Μία άλλη δυνατότητα είναι η αναδιατύπωση, είναι και ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο για την κωδικοποίηση. Θα συμπεριληφθούν στο εφιστάμενο πλαίσιο κάποιες ε, διατάξεις, όμως θα αποσαφινιστούν και ορισμένα κενά με νέες περιπτώσεις. Επίσης, η νομολογία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει με την αναδιατύπωση είναι η εναρμόνιση τομέων που δεν είναι, που δεν βρίσκονται στο εφιστάμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι περιορισμοί, αν και είναι προτιμότερο του πρώτου. Τρίτη πιθανότητα, εναρμόνιση επιλεγμένων ζητημάτων. Για παράδειγμα, τα πνευματικά δικαιώματα δεν είναι εναρμονισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα δικαιώματα των ε, δημιουργών, δικαίωμα προσαρμογής σε προγράμματα τα οποία έχουν ήδη κατοχυρώσει τα πνευματικά τους δικαιώματα. Και η τελευταία επιλογή, να υπάρχει ένας ε, ευρωπαϊκός ε, τίτλος πνευματικών δικαιωμάτων, ο οποίος θα αντικαταστήσει τους εθνικούς και αυτό θα επιφέρει και πλήρη εναρμόνιση. Αυτό θα είναι ένας συνδυασμός των ε, τριών πρώτων επιλογών και θεωρούμε πως ε, θα επιφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. And on side... Ωραία. Και τώρα, για τη δεύτερη ενημέρωση, για τις πτυχές της εσωτερικής αγοράς, να σας εξοικονομήσω λίγο χρόνο, διότι εξήγησα λίγο ποια ήταν τα προβλήματα. Αυτά τα οποία έχουν σημασία για τις πτυχές της εσωτερικής αγοράς είναι κυρίως αυτά τα δύο η κυριαρχία των εδαφικών ε, αδειών και ε, η εδαφικότητα γενικότερα των πνευματικών δικαιωμάτων και οι εξαιρέσει και περιορισμοί για τα πνευματικά δικαιώματα τα οποία ποικίλουν ε, μεταξύ των 28 κρατών μελών. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς στο έκθεση, στο ενημερωτικό σημείωμα, είναι να εξετάζουμε διάφορες επιλογές όπως συνήθως υπάρχει μια επιλογή, μηδενική επιλογή που σημαίνει να μην υπάρξει καμία δράση, ε, μια προσέγγιση ήπιας νομοθεσίας, ε, μια πιο συνολική προσέγγιση με δύο διαφορετικές πτυχές και η ε, τρίτη επιλογή του να χρησιμοποιήσουμε, ε, ε, να έχουμε κάποιες νομοθετικές παρεμβάσεις και να έχουμε και κάποιους τίτλους. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο τον Ανδρέα για να μας παρουσιάσει λίγο τα θέματα αυτά. Η εναρμόνιση των πνευματικών δικαιωμάτων είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία, παρά το γεγονό ότι μπορεί να μην γίνεται και τίποτα για το πλαίσιο αυτό. Η εναρμόνιση θα συνεχιστεί όπω τονίστηκε και στην παρουσίαση του Ανδρέα. Υπάρχει νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που απλώ συμπληρώνει κάποια κενά και ε, ορισμένες φορές με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να έχουμε όλο ένα και πιο εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα υπάρχουν τουλάχιστον δύο νομοθετήματα των οποίων οι συνέπειες πρέπει να αξιολογηθούν και χρειάζεται χρόνος φυσικά, διότι όσον αφορά την ε, οδηγία διαχείρισης των ε, συλλογικών δικαιωμάτων, έχουμε χρόνο μέχρι την άνοιξη του 2016 ε, τα κράτη-μέλη για να εγκρίνουν τη σχετική νομοθεσία και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε πώς η οδηγία αυτή θα επηρεάσει το θέμα της δυνατότητας πολλαπλών αδειών σε διάφορες περιοχές όσον αφορά την επιλογή τη ήπια νομοθεσία, Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση. Ε, έχουν υπάρξει παραδείγματα στα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ε, νομοθέτης, ως αυτός ο οποίος χαράζει μάλλον πολιτική, προσπαθεί να εφαρμόσει μια τέτοια ήπια νομοθεσία και βοηθά απλώς τα κράτη-μέλη και τους ενδιαφερομένους να εγκρίνουν συγκεκριμένε λύσεις οι οποίες δεν θα απατούν καμία νομοθετική παρέμβαση, καμία νομοθετική τροποποίηση παραδείγματο χάρη τη παρεμβάση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στον τομέα τη λογική διαχείριση με μια σύσταση του 2005 που ξεκίνησε μια διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε με την έγκριση τη οδηγία του 2013 επειδή θεωρήθηκε ότι δεν ήταν ικανοποιημένα τα αποτελέσματα τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Θα θυμάστε επίση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια διαδικασία διαμεσολάβηση ε, για τα τέλη και του δασμού σε ε, ιδιωτικά δικαιώματα με βάση την εθνική νομοθεσία και τα προσκόμματα που δημιουργήσει στην εσωτερική αγορά. Εάν αυτές οι επιλογές δεν θεωρηθούν ικανοποιητικές, υπάρχει η νομοθετική δυνατότητα που ε, ανέφεραν και προηγουμένως οι συνάδελφοι. Θεωρούμε ότι υπάρχουν αρκετές δυνατότητες και αυτό γράφουμε και στην έκθεσή μας. Παραδείγματο χάρη, υπάρχει δυνατότητα να στοχεύσουμε συγκεκριμένα και με λεπτομέρεια στο θέμα του κατακαιρματισμού από εξαφική σκοπιά, το θέμα της εδοφικότητα των πνευματικών δικαιωμάτων. Ίσως αυτό θα μπορούσε να υπάρχει δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε μια διάταξη η οποία θα διευκρινίσει βάσει ποιων προϋποθέσεων οι κάτοχοι των δικαιωμάτων μπορούν να λάβουν άδεια ή να δίνουν άδεια συγγνώμη για το έργο τους χώρα χωρίς να παραβιάζουν τη συνθήκη. Αυτό το οποίο έχει προκύψει από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι ότι υπάρχει μία ένταση μεταξύ της εκμετάλλευση των πνευματικών δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο, όπως επιτρέπει η συνθήκη, διότι υπάρχει το άρθρο 36 ότι λέει, που λέει ότι η προστασία τη πνευματική ιδιοκτησία είναι εξαίρεση στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και προσώπων και έχει προκύψει μετά από την απόφαση ε, του δικαστηρίου για την Premier League ότι ε, μπορεί να γίνουν συμβατά με την ιδέα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς που είναι κάτι το οποίο προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ιδιαίτερα. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο εξετάζουμε και περιλαμβάνεται και στην έκθεσή μου είναι η αρχή της χώρας καταγωγής που έχει ήδη συμπεριληφθεί σε συγκεκριμένες οδηγίες. Όπως για παράδειγμα την οδηγία για την ε, μετάδοση έργου το οποίο ε, καλύπτει τα πνευματικά δικαιώματα μέσω δορυφόρων και επίσης ε, την οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα. Όποτε υπάρχει διαδικτυακή μετάδοση, μπορεί η μετάδοση αυτή να υπόκειται απλώς σε ένα νόμο. Δηλαδή, τα δικαιώματα τα οποία ισχύουν σε ένα κράτος μέλος αρκούν για τη διαδικτυακή μετάδοση και μπορεί να γίνει πανευρωπαϊκή διαδικτυακή μετάδοση. Τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, αναφέρθηκε ε, η ιδέα ενός ενωσιακού τίτλου πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι το πιο φιλόδοξο και το πιο ικανοποιητικό μέτρο που θα μπορούσε να ληφθεί από νομοθετική σκοπιά. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει συνένεση μεταξύ των κυβερνήσεων, των κρατών μελών και των νομοθετών ότι χρειάζεται να ενοποιηθεί η νομοθεσία. Διότι όπως ακούστηκε η νομοθεσία αυτή αυτόματα θα υποκαθιστά τα εθνικά ε, μέτρα και τα εθνικά καθεστώτα για τα πνευματικά δικαιώματα. Ε, η ιδέα λοιπόν ότι αυτή η ενιαία ομοσπονδιακή λύση ευρωπαϊκού συστήματος πνευματικών δικαιωμάτων θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί μέσω ενός συστήματος καταχώρησης που θα έχει και συμβατότητα με το διεθνές πλαίσιο για τα ε, πνευματικά δικαιώματα. Το σκεπτικό είναι ότι όπως ε, συμβαίνει και με άλλα δικαιώματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα πνευματικά δικαιώματα, το ευρωπαϊκό επίπεδο προστασίας μπορεί να ενεργοποιείται μέσω ενός συστήματος καταχώρησης. Γνωρίζουμε βέβαια ότι η διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων δεν επιτρέπει να υπάρχει καμία τυπική διαδικασία προκειμένου να εκχωρούνται αυτά τα δικαιώματα, αλλά εμείς θέλουμε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και την εθνική προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, παραδείγματο χάρη οι εθνικέ κινηματογραφικές ταινίες, που μας ενδιαφέρουν σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά επίσης θέλουμε να δώσουμε και τη δυνατότητα στα δικαστήρια να, ε, ε, να εκδίδουν αποφάσεις που θα περιλαμβάνουν πανευρωπαϊκά μέτρα. Ευχαριστώ. Η τέταρτη παρουσίαση τώρα. Okay, I'm Martin Jensen, principal. Είμαι στο VVA εγώ. Είμαι βασικός συνεργάτης Τώρα ετοιμάζουμε το κείμενό μας. Ποιοι είναι οι στόχοι. Να βρούμε ποια είναι τα κενά στην ε, υπάρχουσα νομοθεσία με βάση και τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις να δούμε ποιες ε, λύσεις εναλλακτικές υπάρχουν και μετά κάνουμε μια, μια αποτίμηση αυτών των εναλλακτικών λύσεων και θέλουμε την οικονομική και κοινωνική προστιθέμενη αξία για τους βασικούς παίκτες της ε, εταιρείε διανομής, παραγωγής, τους δημιουργούς, τους ερμηνευτές, τους διαφημιστές και ίσως και τους ε, καταναλωτές. Ποια είναι η μεθοδολογία μας. Πρώτα προσπαθούμε να διαπιστώσουμε τα κενά. Πολλά έχουν υποθεί. Μετά κάνουμε συνεντεύξεις ε, και κάνουμε και μελέτη κειμένων και έχουμε και τους εμπειρογνώμονες. Κάνουμε μια αποτίμηση των εναλλακτικών λύσεων πολιτικής και κάνουμε και ανάλυση κόστους οφέλους. Έχουμε πολλά ποιοτικά στοιχεία που συλλέγει η Κομισιόν μέσω διαβούλευσης με τους εμπλεκομένους φορείς, αλλά έχουμε περιορισμούς για τις διαδικασίες παράβασης και για τις ε, συμβατικές ρυθμίσεις. Οπότε αυτό περιορίζει και την ανάλυση κόστους φέλλου. Ποιοι είναι οι ενωσιακοί στόχοι πολιτικής, για παράδειγμα, σωστό ανταγωνισμό και αμοιβή, σεβασμό θεμελιδών δικαιωμάτων, να προωθήσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση στο δημιουργικό κλάδο και να προωθήσουμε και να προστατεύσουμε τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. Οι δημιουργικές δραστηριότητες είναι γύρω στο 4% του ΑΕΠ της Ένωσης και γύρω στο 3,3% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού εργάζεται σε αυτό τον κλάδο. Σημαντικός λοιπόν κλάδος. Ωστόσο, Έχουμε τεχνολογικές εξελίξεις. Έχουμε περισσότερες ε, διαμεθεωριακές ε, επαφές και ανταλλαγή περιεχομένου και έχουμε περάσει από την ιδιοκτησία του περιεχομένου στην πρόσβαση στο περιεχόμενο. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Χρειάζεται εξυγχρονισμό του πλαισίου προστασία των αδικών δικαιωμάτων. Γιατί μάλλον η παλιά οδηγία πλαίσιο ίσως ε, να μην επαρκεί. Η οργάνωσή μας VVA έχει διαπιστώσει δύο βασικά προβλήματα με την ε, οδηγία πλαίσιο. Πρώτον, η εφαρμογή των πνευματικών δικαιωμάτων διότι δεν υπάρχει σαφήνεια και δεν είναι συμβατή η οδηγία Infosoc και άλλα, με άλλα νομοθετήματα και το δεύτερο δεν υπάρχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για την σωστή αμοιβή για τους ε, δημιουργούς και ερμηνευτές. Τώρα γενικότερα για τον κλάδο. δεν υπάρχει επαρκή συναρμόνιση των κανόνων οπότε η εφαρμογή του πλαισίου σε ενωσιακό επίπεδο δεν είναι πολύ καλή. Θα δούμε θέματα λοιπόν πώς εφαρμόζεται η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και η ισορροπία μεταξύ αυτού και της ελευθερίας πρόσβασης στην πληροφόρηση. Για παράδειγμα, ο περιορισμός σε γεωγραφικές περιοχές. Το geo-blocking, συγκεκριμένου περιεχομένου. Να είναι προσβάσιμο μόνο λοιπόν από ορισμένε ε, γεωγραφικές ζώνες. Το κόστος που αυτό σημαίνει για τις εταιρείε που ε, μεταδίδουν περιεχόμενο, όταν θέλουν να περιορίσουν ε, τη μετάδοσή τους, υπάρχουν διάφοροι κανόνες, κώδικες διοντολογίες Θεωρούμε ότι αν είναι εθελούσαν το τέτοιο σχήμα θα είναι περιορισμένης αποδοτικότητας ενώ αν υπάρχει ένα σύστημα πραγματικά διαμεθοριακής εφαρμογής των πνευματικών δικαιωμάτων και προστασίας τους θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Τέλος, για τη σωστή αμοιβή και αποζημίωση των κατόχων των δικαιωμάτων είναι πολύ διαφορετικές οι καταστάσεις από κλάδο σε κλάδο Άρα έλλειψη διαφάνειας, αφήνειας για τα συμβόλαια σε διάφορους τομείς ή υποτομείς του πολιτιστικού κλάδου. Τέλος, μεγάλες διαφορές μεταξύ των νομικών πλαισίων, των κρατών μελών, για τα συμβόλαια των ε, δημιουργών και ερμηνευτών. Αυτά τα θέματα θα αντιμετωπίσουμε στο κείμενό μας για να υπάρξει ε, σωστή και επαρκής αμοιβή των δημιουργών, των κατόχων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ όλους τους ε, καλεσμένους από την Υπηρεσία Ερευνών για αυτήν την πρώτη γεύση που μας δώσατε για το τι θα περιλαμβάνει η έκθεση και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων όταν δημοσιευθεί η έκθεση. Κύριε Ρέντα, θέλετε να σχολιάσετε. Καταρχάς, ναι, ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Είμαι σίγουρη πως τα τελικά αποτελέσματα θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στην μεταρρύθμιση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η έκθεση που εγκρίναμε σήμερα το πρωί περιέχει πάρα πολλέ συστάσει ε, στο θέμα των εξαιρέσεων και των περιορισμών. Όμω δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε στα αποκλειστικά δικαιώματα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σα ρωτήσω για περισσότερε πληροφορίε σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγή στην ψηφιακή εποχή. Και αν κατάλαβα καλά, υπάρχει ένα θέμα με την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών και τα δικαιώματα τα αναπαραγωγής θα πρέπει να έχουν αποσαφινιστεί. Ποια είναι τα προβλήματα λοιπόν που εντοπίσατε σε αυτόν τον τομέα. Ο κύριος Κάστερ. Καταρχά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις πολύ ενδιαφέρουσε παρουσιάσει. Να πω ότι τονίσατε πως χρειάζεται ένα ξεκάθαρο νομικό ε, πλαίσιο, το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για την αποζημίωση των ε, πολιτισμικών αυτών ε, αγαθών. Τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει διάφορες εξελίξεις, ιδιαίτερα στα πλαίσια τη αξί, της αξίας των ψηφιακό κόσμο. Ιδιαίτερα παρατηρήσαμε ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες ήταν οι κερδισμένοι και οι δημιουργοί ήταν οι χαμένοι. Η πνευματική ιδιοκτησία είναι άραγε το κατάλληλο όργανο για να γίνει αυτή η αναδιανομή του, των κερδών από την πνευματική δημιουργία ή μπορούμε να βρούμε κάποιον άλλο ε, τρόπο. Η πρώτη καποιον αλλο ήταν αυτή. Έπειτα, σε σχέση με την ε, τακτική που θα ακολουθήσουμε για αυτήν την ε, μεταρρύθμιση στην Ευρώπη. Πρέπει άραγε να, να ακολουθήσουμε μια ολιστική προσέγγιση ή να καταπιαστούμε με τους ε, συγκεκριμένους τομείς των πνευματικών δικαιωμάτων, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, τα συγκεκριμένα προβλήματα και να τα λύσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ να απαντήσετε πολύ σύντομα τις ερωτήσεις αυτές, διότι σίγουρα θα έχουμε και αργότερα τη δυνατότητα να τις συζητήσουμε διεξοδικώς. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία Ρέντα σχετικά με την εναρμόνιση των αποκλειστικών δικαιωμάτων. Στη μελέτη μας λάβαμε υπόψη, όπως είπε και η κυρία Ρέντα, τους στόχους της οδηγίας. Και οι στόχοι της οδηγίας σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα έχουν όσο και το πλήστον επιτευχθεί. Λείπουν κάποιες επιπρόσθετες ε, αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράδειγμα. Σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιητική η εναρμόνιση και το επίπεδο αυτής θα μπορούσα να πω. Επίσης, Πραγματικά συμφωνούμε για το ότι υπάρχει μια ασάφεια στο κείμενο σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των ε, ε, πνευματικών ε, δικαιωμάτων έργων που βρίσκονται στην διάθεση του κοινού. Όπως αναφέρατε, δεν υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή νομοθεσία που να αναφέρει αυτόν τον όρο που είπατε. Αυτός ο όρος εφευρέθηκε για να περιγράψει τις επιγραμμικές μεταδόσεις και δεν ήταν επαρκής ε, δυστυχώς για αυτές και μάλιστα σε σημείο που και η επικοινωνία με το κοινό και η αναπαραγωγή θα πρέπει να ε, αποσαφενιστούν έτσι ώστε να δούμε πού βρισκόμαστε νομικά. Είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα και είναι ένα θέμα το οποίο ε, έχει υποστεί μεγάλες απώλειες οικονομικές από την πειρατεία. Είναι ξεχωριστή οντότητα. Γι' αυτό λοιπόν τι σημαίνει ότι υπάρχει κόστος συναλλαγών για την μετάδοση των ε, έργων αυτών που έχουν κατοχυρώσει πνευματική ιδιοκτησία επιγραμμικά. Και δυστυχώς η οδηγία για τη συλλογική διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων δεν καλύπτει αυτούς τους τομείς και θα συνεχίσουμε λοιπόν να έχουμε πρόβλημα εκτός και αν ε, γίνει κάποια νομική, νομοθετική μάλλον παρέμβαση. Και σίγουρα ιδανικά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μπορούσε να εκδώσει μία απόφαση όπου τα δικαιώματα της αναπαραγωγής θα ενσωματωθούν και δεν θα χρειάζεται πλέον να υπάρχει αυτό το επιπρόσθετο κόστος. Όμως δεν έχει ερμηνευτεί έτσι το θέμα αυτό ούτε από το δικαστήριο ούτε από τους ενδιαφερομένους φορείς. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να αντιδράσω στην ερώτηση του κύριου Κιώστερ. Ένα σύντομο σχόλιο σχετικά με τους ε, μεσάζοντες και τους ε, δημιουργούς. Και μετά θα ήθελα να σχολιάσω και αυτήν την ολιστική προσέγγιση που αναφέρατε. Καταρχάς να πω ότι συμφωνώ με τον τρόπο παρουσίασης του προβλήματος αυτού. Τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει μια σταδιακή ενσωμάτωση, αν θέλετε, εντό του, των ε, κερδών από αυτούς τους ε, μεσάζοντες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα λύσει από μόνη της η μεταρρύθμιση του, της Ενωμοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα. Είναι ένα θέμα το οποίο, με το οποίο ασχολείται και η ΓΑΜΑΔΕΛΤΑΚΟΜ για την ψηφιακή αγορά και άλλες υπηρεσίες. Έπειτα η μελέτη αυτή αμφισβητεί τον ε, ρόλο και τη χρησιμότητα αυτών ε, των ε, μέσα ζωντών, ιδιαίτερα στην περίπτωση που έχουν, ιδιαίτερα μάλλον επειδή έχουν κερδίσει πάρα πολλά χρήματα από αυτή τους την δραστηριότητα. Εξετάζουμε λοιπόν το ενδεχόμενο Ενισχυμένη ευθύνη ή ενισχυμένη συνεργασία ανάμεσα στις ε, διαφορετικές αρχές για την επιβολή της ε, νομοθεσίας ή αύξηση της ε, έκθεση στο κοινό ή την αύξηση της αποζημίωσης των δημιουργών. Και εδώ θα απαντήσω και στη δεύτερη ερώτηση, γιατί θα πω ότι είναι ακριβώς η ερώτηση που δεν μπορώ να απαντήσω. Όπως είδατε, έχουμε δύο είδων προτάσεις. Η μία είναι μια εύκολη και γρήγορη λύση, δηλαδή προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν σε τομείς που έχουμε ήδη εντοπίσει και η άλλη πρόταση είναι πιο φιλόδοξη, είναι μια ολιστική προσέγγιση όπου προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια γενικότερη ε, βελτίωση και έναν καλύτερο συνδυασμό όλων των, ε, ε, των πτυχών στην νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε πως η απάντησή μου θα είναι πάρα πολύ προσεκτική. Ναι, μεν υπάρχουν αυτές οι δύο προτάσεις και η πρώτη πρόταση η γρήγορη λύση, δηλαδή λύνη αμέσως τα προβλήματα, όμως μια ολιστική προσέγγιση θα δώσει τις απαντήσεις σε βάθος χρόνου. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας, ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν με το σημείο 27. Και έχουμε ένα περίσσευμα από το πρωί. Το σημείο 24 της κυρίας Κάουφμαν. εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Ο λόγος στην κυρία Κάφμαν. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή έχει περάσει η ώρα, θα προσπαθήσω να μην μακρηγορήσω. Κάναμε ήδη μια συζήτηση και το κείμενο της γνωμοδότησής μου το έχετε λάβει. Πρέπει να πω ότι για μένα είναι σημαντικό να κάνουμε όλοι μαζί ό,τι μπορούμε, ώστε αυτό το μέσο Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών να βελτιωθεί ουσιαστικά, να είναι πιο φιλική προς τον χρήστη. Διότι δυστυχώς υπευλήθησαν 51 τέτοιες πρωτοβουλίες Οι 20 δεν έγιναν αποδεκτές. Οι 31 θεωρήθησαν αποδεκτές. Αλλά μόνον τρεις λοιπόν συνολικά επέτυχαν τον αναγκαίο αριθμό υπογραφών. Άρα πρέπει όλοι να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε μια σειρά από γραφειοκρατικούς φραγμούς που είναι ακόμη στον κανονισμό. Αυτός είναι ο στόχος και του συναδέλφου Σέπλη που είναι εισηγητής στην ΑΦΚΟ. Ποια σημεία θεωρώ πολύ σημαντικά. Εν παρόδο, ανέλαβα να ασχοληθώ με το θέμα αυτό γιατί χαίρομαι πολύ που η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ασχολείται με το θέμα των μεταφράσεων που αφορά τις πρωτοβουλίες αυτές και θα βοηθήσει λοιπόν τις πρωτοβουλίες. Τώρα, επανέρχομαι στον κανονισμό. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ενιαίες απαιτήσει για τα προσωπικά στοιχεία. Στόχος μας να απλοποιήσουμε τη διαδικασία συλλογής υπογραφών και πρέπει επίσης να τονίσουμε να καταργήσουμε την ανάγκη συμπερίληψης του αριθμού ταυτότητας των υπογραφών όπως λέει το σημείο 6. Πολύ συχνά όμως η Κομισιόν δεν κάνει δεκτές αυτές τις πρωτοβουλίες λέγοντας ότι είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια άλλη διαδικασία, να υποστηρίζουμε αυτούς που ε, αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία, να υπάρξει μια πρωτοβουλία, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε. γιατί υπάρχουν λεπτά θέματα, ε, πολύ περίπλοκα. Τι ακριβώς ε, μπορεί να γίνει παραδεκτό, τι νομικά είναι εντός των αρμοδιοτήτων. Στο σημείο 7, όπως θα θυμάστε, την προηγούμενη φορά που το συζητήσαμε, είχαμε πει ότι πολλοί διαμαρτύρονται ότι η δωδεκάμινη περίοδος συλλογής υπογραφών είναι περιορισμένη. και επίσης διαμαρτύρονται αυτοί που ανέλαβαν την, ε, ε, την πρωτοβουλία λένε ότι έχει πολύ οργανωτική δουλειά λοιπόν αυτό θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τον κανονισμό και να καταργήσουμε αυτή την αυτόματη σύνδεση που υπάρχει τώρα στον κανονισμό ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία των πολιτών έχει μόνο 12 μήνες από τη στιγμή που η Κομισιόν την εγγράφει. Αν μπορούμε να τα αποσυνδέσουμε αυτά τα δύο, τότε θα μπορούσαν να αποφασίζουν οι ίδιοι που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία από ποια στιγμή και πέρα θα αρχίσουν να συλλέγουν υπογραφέ, από τη στιγμή που έχουν δηλαδή προετοιμαστεί επαρκώ και τότε θα επαρκούσε το 12 μήνο. Ε, παρακαλώ όλους τους αδέλφους να υποστηρίξουν το σημείο 9. Είμαι ιδιαιτέρως υπέρ μιας ενιαίας διαδικασίας. Το ότι το συνέσαμε με το ενεργό δικαίωμα ψήφου έχει να κάνει με το ότι στην Αυστρία ακόμη και 16 χρόνια μπορούν να υπογράψουν. Σε όλες τις άλλες χώρες είναι από 18 και πάνω. Πρέπει λοιπόν να απευθυνθούμε προς τους νέους, να τους πλησιάσουμε να τους στηρίξουμε, να τους βοηθήσουμε να μάθουν για την Ευρώπη, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, να, να το διαχωρίσουμε σαφώς από το δικαίωμα εκλέγην και εκλέγεστε. Ούτως ώστε να μπορούν και οι 16χρονοι παντού να υπογράφουν. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά σημεία που καλό θα ήταν να εγκριθούν ούτω ώστε να γίνει πιο φιλική προς τους πολίτες η διαδικασία αυτή. Πρέπει λοιπόν να αναθεωρηθεί αυτός ο κανονισμός και αυτό είναι το κεντρικό θέμα που αναφέρω στο 11 της γνωμοδότησής μου. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι πολύ περιορισμένη μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 23 τρέχοντος η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα γίνει στις 13-14 Ιουλίου. Πριν λοιπόν τις διακοπές. Και με χαρά να δω τις ε, τροπολογίες των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κάφμαν. Θέλει κανείς το λόγο. Κύριος Κώστα. Ευχαριστώ. Σίλβια για την πολύ καλή ενημέρωση. Τονίζεις ότι αυτή η σημαντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που για μένα είναι σημαντική ούτω ώστε να φέρουν πιο κοντά τους πολίτες με τα θεσμικά όργανα λες ότι πρέπει να είναι πιο φιλική προς το χρήστη αλλά δεν σχετίζεται το ότι δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς με το ότι έχει περιορισμένη δυνατότητα να αλλάξει τα πράγματα Δηλαδή οι πρωτοβουλίε κυρίω απευθύνονται προς την Κομισιόν. Και η Κομισιόν αποφασίζει τι θα κάνει. Μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δεν θα μπορούσε να απευθύνεται απευθεία στο Κοινοβούλιο. Να ασχολείται το Κοινοβούλιο με αυτά. Και το Κοινοβούλιο να αποφασίζει. Μήπω θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω. Να είναι ένα είδος ε, δημοψήφισμα για θέματα συγκεκριμένης ουσίας. Ευχαριστώ κύριος ε, Λιμπερτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν ε, περάσω στην ουσία του ζητήματος, θα ήθελα να αναφερθώ στη σημερινή συνεδρίαση που νομίζω ότι είχε πολύ επιβαρημένη ημερήσια διάταξη. Σήμερα είχαμε τρία πολύ σημαντικά ζητήματα για τα δικαιώματα των δημιουργών ε, και τα υπόλοιπα και χρειάστηκε και εμείς και οι βοηθείς μας να εργαζόμαστε συνεχώς με συμβαστικές τροπολογίε που έφταναν την τελευταία στιγμή στα αγγλικά και θα ήθελα σας παρακαλώ να μην ξανασυμβεί αυτό. Από εδώ και πέρα να είναι λίγο πιο ελαφριά η μερίσια διάταξη. επειδή θα υπάρξει και μία ε, νέα επιτροπή, κατά πάσα πιθανότητα θα είμαι μια νέα πολιτική ομάδα ε, θα είμαι μάλλον συντονιστής και θα ήθελα να μην είναι τόσο επιβερημένα τα πράγματα. Τώρα, στο θέμα. Φαίνεται ότι έχουμε παραπλανηθεί οι Ευρωπαίοι πολίτες από αυτό το μηχανισμό. Υπάρχουν μόνο τρία θετικά αποτελέσματα μέχρι τώρα για το θέμα αυτό και είναι πάρα πολύ λίγα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για τους λόγους αυτής της αποτυχίας. όσοι υπάρχουν κάποια συγκυριακά ζητήματα τα οποία αναφέρονται και στην έκθεση και υπάρχουν και θέματα ουσίας τα οποία όμως δεν αναφέρονται στην έκθεση και θα ήθελα να σας τα αναφέρω εδώ. Καταρχάς, οι συγκυριακοί λόγοι ε, έχουν σχέση απλώς και μόνο με το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιες ε, ε, προβληματικές πτυχές από την αρχική ε, σύλληψη της έννοιας αυτής. Παραδείγματο χάρη δεν υπήρχε διακτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρκετά σαφής, το αναφέρει και έκθεση αυτό. Ε, επομένως κάποιοι πολίτες έκανε λάθος, υπάρχουν και κάποια άλλα προβλήματα τα οποία ε, αναφέρονται στην ανάγκη ε, που προέκυψε από κάποια κράτη-μέλη όταν υπογράφεται ε, μία ε, πρόταση από κάποιο πολίτη θα πρέπει να υπάρχει και ένας προσωπικός αριθμός αναγνώρισης ταυτότητας που σημαίνει ότι ήταν μεγάλη επιβάρυνση και ήταν γραφειοκρατικό το ζήτημα για τους πολίτες και επίσης υπάρχουν και κάποιοι άλλοι κανόνες ε, που καταδεικνύουν ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι περίπλοκο, οι κανόνες για τον αριθμό των υπογραφών και τον αριθμό των χωρών από τις οποίες θα πρέπει να προέρχονται οι υπογράφοντες είναι αρκετά περίπλοκοι και αυτό σημαίνει ότι για αυτούς τους λόγους η πρωτοβουλία αυτή ε, ήταν ιδιαίτερα απογοητευτική. Αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Υπάρχουν και λόγοι ουσίας, οι οποίοι έχουν να κάνουν με το μηχανισμό όπως ε, συστάθηκε βάσει το άρθρο 5 της συνθήκης. Χρειάζονται 1 εκατομμύριο πολίτες και αυτή τη στιγμή και από 7 διαφορετικές χώρες μέλη, αλλά το πρόβλημα είναι ότι στο κάτω-κάτω της γραφής πρόκειται για μια πολύ ε, επαχθή διαδικασία που δεν αξίζει τον κόπο διότι τελικά ε, απλώς επιτρέπει στους πολίτες να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να αλλάξει μια νομοθετική πρόταση. Αυτή η πρόσκληση όμως δεν αρκεί. Ε, δεν είναι διατεθειμένοι οι πολίτες να ξεκινήσουν αυτή την επαχθή διαδικασία απλώς και μόνο για μια πρόσκληση. Και υπάρχουν και πολλές αποτυχίες. Για παράδειγμα, η ε, ε, διαβόητη απόπειρα για να σταματήσει το TTIP, ε, τη σταμάτησε αμέσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είπε ότι δεν είναι αποδεκτή. Αν προχωρήσουμε περαιτέρω, θα υπάρξει εδώ μια διαδικασία, η οποία θα είναι μια διαδικασία συμμετοχής του λαού που είναι μια σημαντική επιλογή αλλά δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε τα πράγματα. Δεν είναι μια διαδικασία συμμετοχικής δημοκρατίας αυτή που έχουμε. Η διαδικασία συμμετοχικής, ε, ε, δημοκρατικής... συμμετοχικής δημοκρατίας που αναφέρεται στο σημείο 1 της έκθεσης ε, είναι κάτι άλλο. Η δημοκρατία βάσει των κλασικών ορισμών είναι το δικαίωμα των λαών. Επομένως αυτό θα πρέπει να επιτρέπεται ε, στους πολίτες. Μέσω του νόμου θα πρέπει να έχουν την εξησία να έχουν τον τελευταίο λόγο. Η συμμετοχή δημοκρατία είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Επιτρέπει απλώς, το βλέπουμε εδώ, στο λαό να εκφράσει την άποψή του, να εκφράσει απλώς μία πρόσκληση. Και η πρόσκληση δεν είναι αποφασίζω για την τύχη μου. Εάν λοιπόν πραγματικά θέλουμε να αναζωογονήσουμε αυτή τη διαδικασία της συμμετοχής δημοκρατία θα πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα, να εξηγήσουμε ότι αυτή δεν είναι μια διαδικασία συμμετοχικής δημοκρατίας, είναι κάτι άλλο και από εκεί και πέρα θα πρέπει να αναρωτηθούμε και για τους λόγους για τους οποίους αποθαρρύνουμε τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης, ιδέως ε, ξεκινώντας από το παράδειγμα του Stop TTIP που για μένα είναι ένα παράδειγμα το οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Η κυρία Κάουφμαν θέλει να απαντήσει. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρόλες τις ε, κριτικές ε, που ακούστηκαν, ε, θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι καινούριο. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει διεθνική συμμετοχική δημοκρατία. Η πρωτοβουλία των πολιτών είναι κάτι πρωτοποριακό σε αυτόν τον τομέα. Ε, βρίσκεται, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της συνθήκης της Λισαβόνας και ε, έχει τεθεί σε λειτουργία. Και χαίρομαι πάρα πολύ με το ότι μετά από τρία χρόνια βλέπουμε την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και βλέπουμε τι έχει λειτουργήσει σωστά και ποια προβλήματα υπάρχουν. Και το γεγονός ότι κάποια προβλήματα προέκυψαν δεν σημαίνει ότι πρέπει να αμφισβητήσουμε όλον τον κανονισμό. Και μάλιστα στην ε, γνωμοδότησή μου αναφέρομαι σε κάποια από αυτά προβλήματα. Τώρα η πρωτοβουλία των πολιτών και οι υπογραφές που χρειάζονται, το 1 εκατομμύριο υπογραφών, είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε. Πιστεύω όμως πως δεν χρειάζεται ε, παραπάνω συζήτηση, διότι οι διατάξεις στην συνθήκη είναι ξεκάθαρες. Και να σας υπενθυμίσω ότι αυτές ε, οι διατάξεις χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια για να ενσωματωθούν στις ε, συνθήκες. Ωστόσο αυτό που είναι σαφές είναι ότι εάν θέλουμε να λειτουργεί σωστά η πρωτοβουλία των πολιτών και να υπάρχει η λειτουργία τη ε, της ε, πρωτοβουλίας αυτής, χρειάζονται σαφείς ε, διατάξει και ένα σαφές πλαίσιο. Όπως ερώτησε τώρα και ο, όπως είπε και ο συνάδελφος Κώστερ, δεν μιλάμε για δημοψήφισμα, διότι σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν άλλα μέσα. Στο Βερολίνο, για παράδειγμα, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, γίνονται πάρα πολλά δημοψηφίσματα, τα οποία ακυρώνουν αποφάσεις ε, του τοπικού κοινοβουλίου. Δεν ε, πρόκειται λοιπόν για κάτι τέτοιο. Ε, πρόκειται για την δυνατότητα που θέλουμε να δώσουμε στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής. Να συνδεθούν λοιπόν με τους υπόλοιπους πολίτες στα άλλα κρατημέλη για να δουν τα κοινά που έχουν και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε νομοθετικό επίπεδο για εκείνους. Αυτή λοιπόν η διαδικασία είναι για μένα κάτι πάρα πολύ καλό και ορίζεται, καθορίζεται σαφέστατα στον κανονισμό. Όπου ε, ο κύριο Κώστα έκανε μια πρόταση να απευθύνονται οι πρωτοβουλίε αυτέ στο Κοινοβούλιο. Να σας πω ότι έχουμε την Επιτροπή Αναφορών που κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα με τις αναφορές των πολιτών και οι αναφορές με την πρωτοβουλία των πολιτών είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Για μένα σημαντικό είναι στην πρωτοβουλία των πολιτών ο πολίτης να συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία. Και εάν χρειάζονται ένα εκατομμύριο υπογραφές ε, ή όχι, αυτό μπορούμε να το εξετάσουμε, μπορούμε να διοργανώσουμε μια κρόαση για παράδειγμα, όπως είδαμε και στην τελευταία επιτυχημένη πρωτοβουλία των πολιτών, το σταματήστε τη ζωοτομία. Και βλέπετε λοιπόν ότι όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο της εξέτασης μια τεράστιας πρωτοβουλίας, πόσο διαφορετικές είναι οι απόψεις των πολιτών και ε, πόσο σημαντικό είναι να το γνωρίζουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε αυτή τη δυνατότητα για να μπορέσουμε να ακούσουμε όλες τις απόψεις και να διαμορφώσουμε άποψη και σίγουρα η αλλαγή, η κατάργηση της πρωτοβουλίας των πολιτών δεν είναι ο τρόπος ε, για να το πράξουμε αυτό. Τώρα, αυτός ο αριθμός, το 1 εκατομμύριο των υπογραφών, ιδιαίτερα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με 500 εκατομμύρια κατοίκους είναι ε, πιστεύω αρκετό. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ε, που δεν αφήνει τους πολίτες να αρχίσουν μια δική τους πρωτοβουλία, δεν, δεν, τους εμποδίζει κανείς. Και αυτό το βλέπουμε από τις ε, πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί. Βλέπουμε πως έχουμε υποτιμήσει την ε, δουλειά που έχει γίνει από τους πολίτες μέχρι να φτάσουν σε αυτό το σημείο της συγκέντρωσης ενός εκατομμυρίου υπογραφών. Και βλέπουμε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές χρειάζονται πάρα πολύ δουλειά από το, στάδιο, από το αρχικό στάδιο μέχρι την ε, εξέταση από την Επιτροπή, την διαδικασία διοργανώσεις ακροάσεων. Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ δουλειά. Και χρειάζεται επίσης να αυξήσουμε την ορατότητα του μέσου αυτού, διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ γνωστό, δεν είναι όσο θα έπρεπε γνωστό στην Ευρώπη. Πρέπει να το διαφημίσουμε, έτσι ώστε οι πολίτες να ξέρουν τι δυνατότητες έχουν. Και εδώ πραγματικά μπορώ να πω ότι συνεχίζουμε να υστερούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάουφμαν. Με αυτή την παρέμβασή σας λοιπόν τελειώσαμε με το σημείο 24 και περνάμε τώρα στο σημείο 29, εξέταση των τροπολογιών για την 30η και 31η ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λόγο έχει ο εισηγητής κύριος Χρυσόγονος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής για τις ε, τροπολογίες που υπέβαλαν στο σχέδιο έκθεσης για την παρακολούθηση της εφαρμογής του, της Ευρωπαϊκού Δικαίου από το 2012 στο 2013. Υπάρχουν ενδείξεις του πόσο σοβαρό είναι το θέμα αυτό με τις 60 τροπολογίες και μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνέπειες της Επιτροπής μας και την επιρροή της ε, υποβάλλοντας μια συνολική έκθεση παρά το γεγονός ότι συνάδει με τις αντίστοιχες εκθέσεις ε, για το ίδιο θέμα θα έχει κάποια νέα στοιχεία και ίσως θα λάβει υπόψη της ευρύτερα το ζήτημα το οποίο εξετάζουμε. Έχω ήδη εξετάσει όλες τις τροπολογίες σας. Έχω δει ότι κάποιες εξ αυτών ε, πηγαίνουν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των ιδεών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο έκθεσης, κάποιες είναι αντίθετες σε αυτό το οποίο προτείνεται στο σχέδιο έκθεσης και κάποιες άλλες εισαγάγουν κάποιες νέες προπτικές οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στο σχέδιο. Βεβαίω δεν μπορούμε να συμφωνούμε επί όλων των θεμάτων, αλλά είμαι βέβαιο ότι για τις περισσότερε από τι προτινόμενε τροπολογίε μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να βρούμε κοινό έδαφο. Έχω ξεκινήσει ήδη τις εργασίες για συμβιβαστικέ τροπολογίε, αλλά φυσικά θα ήθελα να ακούσω και τη θέση σα εδώ στην Ευρωπαϊκή ε, ε, στην Επιτροπή μα, και να έχουμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε τι αρδίε και τι προτάσει σα. Έτσι θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα πώ θα πρέπει να αντιληφθούμε τα θέματα τα οποία εξετάζουμε και πώς μπορώ να εργαστώ αποτελεσματικά για να σας παρουσιάσω ένα σύνολο συμβιβαστικών τροπολογιών που στη συνέχεια θα συζητηθούν εις βάθος ε, και σε λεπτομέρειες ε, στη συνεδριάση των σπιωδών εισηγητών. Ως τελευταία παρατήρηση θα ήθελα να πω ότι η πεμπτουσία του σχεδίου έκθεσής μου είναι μια απόπειρα η οποία εδράζεται σε κάποια ίσως δυσάρεστα στοιχεία. Καταρχάς το γεγονός ότι υπάρχει μια διάκριση μεταξύ ε, πρωτογενούς και δευτερεύοντος δικαίου και ορισμένες φορές ε, το δευτερογενές δίκαιο είναι, ε, υπερβαίνει το πρωτεύον δίκαιο. Επίσης, το ευρωπαϊκό δίκαιο μπορεί να προέρχεται όχι μόνο από τα θεσμικά όργανα των κρατών μελών, αλλά και από τα θεσμικά όργανα των κρατών μελών, διότι μπορεί να παραβιάζεται το πρωτεύον δίκαιο και κάποια συγκεκριμένα δικαιώματα μέσω της συμπεριφοράς τους. Οι πολιτικές λιτότητας οι οποίες επευλήθησαν την τελευταία πενταετία ή στα τελευταία έξι χρόνια προκειμένου να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση, ιδίω εντός της Ευρωζώνης, έχουν θέσει πολύ σοβαρούς περιορισμούς, κυρίως στα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, τα οποία είναι εγγεγρωμένα στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό περιγράφεται ήδη ε, στην πολύ αναλυτική και διεξοδική μελέτη για την Γενική Διεύθυνση για τις Εσωτερικές Πολιτικές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που μελετά τις συνέπειες της κρίσης ε, για τα θεμελιώδη δικαιώματα που δημοσιεύθηκε πριν από κάποιες εβδομάδες κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ε, Πολιτικών Ελευθεριών του Κοινοβουλίου και περιλαμβάνεται στο σχέδιο έκθεσής Η άποψή μου ότι μία είναι ότι μία έκθεση που αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου σε χρόνια κρίσης, όπως το 2012 και το 2013, πρέπει να ασχοληθεί με τα προβλήματα αυτά, ώστε να είναι και λίγο πιστικό για τους Ευρωπαίους πολίτες που μπορεί να τη διαβάσουν. Βέβαια, αν το επιθυμεί η πλειοψηφία, η Επιτροπή μας και η Ολομέλεια εν τέλει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσε απλώς να παραγνωρίσει αυτά τα στοιχεία και να διαγράψει οποιαδήποτε αναφορά στη λιτότητα, στα κοινωνικά δικαιώματα και στις προβληματικές σχέσεις τους. Αυτό βέβαια δεν θα επιλύσει τα υφιστάμενα προβλήματα, απλώς θα καταδείξει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αποδεχτεί την πραγματικότητα και δεν μπορεί να προσπαθήσει να τα επιλύσει κατά τρόπον ώστε να βοηθήσει και την ευρωπαϊκή διαδικασία ολοκλήρωσης η οποία θα πρέπει να βασίζεται κυρίως στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Θέλει κάποιος το λόγο. Η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Χρυσόγονο, Χρυσόγονε για το σχέδιο εκθεσής σας, το οποίο ήδη αναφέρθηκε στα φλέγοντα θέματα της έκθεσης, τα θέματα τα οποία δημιουργούν αντιθέσεις εδώ στα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό φυσικά έχει να κάνει με τις συνέπειες ε, λόγω των μέτρων λιτότητας ε, ε, και το γεγονός ότι παραβιάζονται δεσμευτικές ε, συνθήκες ε, συμπεριλαμβανομένου και του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι είναι υγιές να αναγνωρίσουμε τι έχει συμβεί, χωρίς ίσως να πρέπει να επισέλθουμε σε πώς λέει λεπτομέρειες για το πώς μπορούμε να επιλύσουμε την κρίση και τη λιτότητα. Δεν με έχετε πείσει όταν λέτε ότι τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τρόικας έχουν παραβιάσει τα δικαιώματα των κρατών μελών, κυρίως του δικού σας είναι το δικαίωμα των κρατών μελών να επιλέγουν ελεύθερα τον τρόπο της ιδιοκτησίας τους, να αναφέρεστε στις ιδιωτικοποίησεις. Αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν κάπως να αναγνωριστεί ότι τα μέτρα λιτότητας έχουν δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις τις οποίες ε, έχουν παραβιαστεί ε, οι διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Όσον αφορά κάποιες άλλες πτυχές, εδώ θα ήθελα ίσως να τονίσω και κάτι το οποίο έχω υποβάλει και ως τροπολογία. Βάσει του χάρτη, οι πολίτες έχουν δικαίωμα σε χρηστή διοίκηση. Επομένως, θα πρέπει να επαναλάβουμε την έκκλησή μας για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις Διοικητικές Διαδικασίες γεγονός το οποίο θα επιτρέψει στους πολίτες να έχουν εφαρμογή αυτού του δικαιώματος. Να σας υπενθυμίσω ότι η νομική βάση στη συνθήκη της Λισαβόνα, το άρθρο 298, είναι το μόνο άρθρο, η μόνη νομική βάση που μέχρι τούδε δεν έχει εφαρμοστεί. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι λοιπόν για τον νόμο για τις διοικητικές διαδικασίες. Όσον αφορά τις διαδικασίες επί παραβάση τώρα, ε, από το σχέδιο εκθεσής σας ε, διαπιστώνω με ενδιαφέρον ότι ο αριθμός ε, των παραβιάσεων για τη μεταφορά έχει μειωθεί και από την έκθεση αναφέρεται ότι κάποια εργαλεία όπως το EU Pilot έχουν βοηθήσει. Θα ήθελα να συμπεριλάβουμε και την παρατήρηση ότι το EU Pilot δεν νομιμοποιείται και πρέπει να γίνει μιας κάποιας μορφής νομικά δεσμευτικό εργαλείο που θα περιλαμβάνει τις διάφορες διαδικασίες, τα διάφορα στάδια των διαδικασιών επί παραβάση. Ίσως αυτό θα μπορούσαμε να το λάβουμε υπόψη. Τώρα, το gold plating, αυτή η υπερβολική νομοθεσία και διαδικασία σε εθνικό επίπεδο. Ε, αναφέρεται σε κάποιες τροπολογίες, ίσως δεν ήταν στην έκθεσή σας. Ίσως καλό θα ήταν να υπενθυμίζουμε στα κράτη-μέλη όταν μεταφέρουν εθνική νομοθεσία ότι ε, σχεδόν τείνουν να κρύβουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν απορρέουν από τα ευρωπαϊκά νομικά μέσα. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια τουλάχιστον και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να κάνουν διάκριση μεταξύ των υποχρεώσεων τους να μεταφέρουν κάτι αφενός και αφετέρου κάποια άλλα στοιχεία τα οποία θεωρούν ότι είναι απαραίτητα να προσθέσουν. Μου αρέσει η τροπολογία του κυρίου Κάριμ και άλλων, η παριθμό 57, που υποστηρίζει το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην μεταφορά του ευρωπαϊκού δικαίου. Ορισμένες φορές θεωρώ ότι οι ανταλλαγέ απόψεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων δεν είναι πάντα χρήσιμοι, αλλά όταν είναι χρήσιμοι είναι γιατί γίνεται μια ανταλλαγή εμπειριών για ποιο λόγο πρέπει να μεταφερθούν τα συγκεκριμένα μέσα. Και να αναφερθώ και σε κάτι που δεν έχει ίσως ε, σχέση με την έκθεση, αλλά υπάρχουν τρεις χώρες που έχουν συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Γεωργία. Και οι χώρες αυτές υποχρεούνται να μεταφέρουν 300 με 400 νομοθετικά μέσα, ε, συμπεριλαμβανόμενων και ο κανόνων για την εσωτερική αγορά, τις δημόσιες συμβάσεις, όλα τα δύσκολα. Και ίσως θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να βοηθήσει αυτές τις χώρες, τα εθνικά τους κοινοβούλια, να κάνουν μεταφορά της συγκεκριμένη νομοθεσία. Ελπίζουμε να έχουμε κάτι καλό από την εκθεσή σας και ίσως ε, ε, οι συνάδελφοι θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι τα μέτρα λιτότητας όντως έχουν παραβιάσει κάποιες ε, αρχές και κανόνες του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο Le, rapport de monsieur... Η έκθεση του κυρίου Χρυσόγονου είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει μια αρετή. Δεν μιλάει ξύλινη γλώσσα. Υπογραμμίζει ότι είναι η άποψή του και η δική μου, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της κρίσης, υποχρέωσε τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν τις χέρες να παραβιάσουν θεμελιώδη δικαιώματα και το χάρτη, τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης, σωστό, Σκεφτόμαστε φυσικά διαβάζοντας το παράδειγμα της Ελλάδας, όπου η πρόσβαση για παράδειγμα στην ε, περίθαλψη έχει φύγει, γιατί δυστυχώς έχει ανέβει η παιδική και ευρεφική θνησιμότητα και το δικαίωμα στην κατοικία κινδυνεύει σε πολλές χώρες στην Ευρώπη. Λυπάμαι ωστόσο, ε, διαβάζοντας τις τροπολογίες που διαπιστώνω, ότι όλα αυτά τα τμήματα που απεκάλυπταν αυτή την αλήθεια με πολύ σαφή τρόπο θα διαγραφούν. Τα σημεία 7, 8, 9, τα ιετολογικές σκέψεις F και G δεν θα αντισταθούν στη τρόπο τροπολογιών. Θα επανέλθουμε λοιπόν στην συνήθι ξύλινη γλώσσα και τελικά θα παραχθεί ένα κείμενο που διαβάζοντάς το θα καταλήγουμε σε λάθος συμπεράσματα. Δεν είμαστε σε θέση να πούμε τα πράγματα στα ράτα. Ένα στοιχείο είναι πολύ ενδιαφέρον που αποκαλύπτει η έκθεση. Μια ανάλυση της Κομισιόν που είναι ιδιαίτερα κοινική. Παραθέτω, η Κομισιόν ε, θεωρεί ότι τα πρωτόκολλα οικονομικής προσέγγισης δεν είναι νομοθετικά κείμενα της Ένωσης και άρα δεν ισχύει για αυτά ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι απαράδεκτο αυτό διότι αιτιολογεί και δικαιολογεί την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για να πω κάτι πιο ευχάριστο καταληκτικά, ορισμένες τροπολογίες είναι ενδιαφέρουσες. Μία που στηρίζω σίγουρα είναι η 27 της κυρίας Χάουταλα που προτείνει να διευκρινίσουμε το νομικό καθεστώς του EU Pilot. Αυτό είναι καλή ιδέα. Είναι ένας οργανισμός που παρεμβαίνει λοιπόν στον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης Πρέπει λοιπόν να διευκρινιστεί, να καταλάβουμε και οι πολίτες να καταλάβουν τι ρόλο παίζει αυτός ο φορέας και πώς ακριβώς παρεμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καστάλτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο συζητητής στην Επιτροπή ΑΦΚΟ της γνωμοδότησης ήθελα να είμαι παρόν για να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Χρυσόγονο, για τη δουλειά του. Οι παρατήρησει μου θα είναι μάλλον τεχνικού χαρακτήρα και θα σταθώ στα σημεία 3, 4, 5 και 6, τα οποία είναι και θέματα της ε, αρμοδιότητας της δικής μου επιτροπής. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι συμφωνούμε απόλυτα στα πολιτικά σημεία τα οποία εκφράζει η έκθεση, τα σημεία ρήξης που επισημαίνουν ότι οι πολιτικές λιτότητες έχουν γονατίσει και έχουν διακυβευτεί δικαιώματα τα οποία θα έπρεπε να είναι αναφέρετα δικαιώματα όλων των Ευρωπαίων πολιτών και βλέπουμε από την πραγματικότητα ότι ε, λησμονούνται και παραγωνίζονται για να μην πω ότι τους ταρνούνται και σε κάποιες περιπτώσεις στις χώρες της Μεσογείου ε, και αφήνουμε τους ανθρώπους στη μοίρα τους. Όσον αφορά το σημείο 3, Σαφώς και εμείς στην Επιτροπή ΑΦΚΟ επισημάναμε τη σημασία μιας πιθανής κύρωσης από την πρώτη καταδίκη ε, μη τήρησης της νομοθεσίας και εδώ συμφωνούμε. Όσον αφορά το σημείο 4, νομίζω ότι αυτό το ανέφεραν και οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από μένα υπήρξε και μια αντιπαράθεση μεταξύ των συναδέλφων των διαφέρων ομάδων και τελικώς ε, όλοι συμφωνήσαμε στο γεγονός ότι επειδή δεν υπάρχει ε, νομικό καθεστώς για το EU Pilot, δεδομένου ότι είναι ένας μηχανισμός συνεργασίας και δεν έχει ε, θεσμοθετηθεί πλήρως, το ενδεχόμενο να υπάρχει μια διακριτική ευχέρεια για τις διάφορες επιτροπές δεν επιτρέπει να έχουμε τις προδιαγραφές διαφάνειας και λογοδοσίας που θα έπρεπε να υπάρχουν σε αυτό το μηχανισμό. Επομένως υποστηρίζουμε πλήρως αυτό που έλεγε και η συνάδελφος Χάουταλα προηγουμένως όσον αφορά το νομικό καθεστώς του και επίσης ε, ε, έχουμε πιέσει ώστε να υπάρχει ένα αυτόνομο σύστημα αξιολόγησης μετά ε, την, ε, ε, την εφαρμογή σε εσωτερικό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να υπάρχει ένας υποχρεωτικός πίνακας αντιστοιχίας για να φανεί πόσο σημαντικό είναι, με, ειδικά μετά από τη διαδικασία της Λισαβόνας, εμείς ως νομοθέτες να προσδώσουμε διαφάνεια και αναγνωρισιμότητα στην αξιολόγηση και την εφαρμογή από πλευράς κρατών μελών. Όσον αφορά το σημείο 5, το οποίο συνδέεται εν μέρη και με αυτό που έλεγα προηγουμένως για την πολιτική αξιολόγηση, οι πολίτες πρέπει να είναι απόλυτα βέβαιοι, ε, να γνωρίζουν ότι λειτουργεί το δίκαιο και αυτό θα πρέπει να είναι και η πρώτη μας μέρημνα και πολύ καλά επισημαίνεται εδώ στην έκθεση. Τέλος, όσον αφορά το σημείο 6 και την ευθύνη για την εφαρμογή της ε, ε, Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στα κράτη-μέλη, σταθήκαμε πάρα πολύ και στην ανάγκη να αποφύγουμε το gold plating και οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην γίνονται αντιληπτοί με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο καθής. Ελπίζω όλες οι προτάσεις μας ε, και όσα αναφέρονται στη γνωμοδότησή μας να γίνουν δεκτά και να ληφθούν, υπόψη από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Σας ευχαριστώ. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο τελευταίος ομιλητής. Κύριε Χρυσόγονε, θέλετε να αντιδράσετε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους και προσβλέπω στην συνεργασία στα πλαίσια της ε, συνάντησης των σκιωδών για να βρούμε τους συμβασμούς όπου μπορούμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Οπότε κλείνουμε και αυτό το θέμα. Και περνάμε στο 31. Ανταλλαγή απόψεων. Για την ε, πράξη για τη διασυνδεδεμένη ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά. Ο κύριος Τσαμπάσκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε χαρά μου να είμαι εισηγητής για ένα τόσο σημαντικό θέμα και ξεκινάω με ανυπομονησία την εργασία μου. Είχαμε μια ανταλλαγή σήμερα με τους σκιώδεις. Είχαμε προβλέψει και μια άλλη αύριο. Η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά που πρότεινε η Κομισιόν αρχές Μαΐου έχει στόχο να προσφέρει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις αυξημένες δυνατότητες ανάπτυξης στα πλαίσια των ψηφιακών υπηρεσιών. Αυτή η στρατηγική ε, καταλήγει σε μια σειρά από πρωτοβουλίες που είναι αρμοδιότητα διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Στο σχέδιο γνωμοδότησης εστιάζω στα θέματα που είναι αρμοδιότητα τη δική μας επιτροπής. Ιδιαίτερα αφορά το ρόλο της ψηφιακής αγοράς στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης, της καινοτομίας, το δημιουργικό τομέα, στην ανταγωνιστικότητα, καταργώντας ε, τους υπάρχοντες φραγμούς, την ανάγκη μεταρρυθμίσεων για να βελτιώσουμε την φορητότητα των περιεχομένων που ε, νομίμως μπορεί να μεταφέρει κανείς να βελτιώσουμε τις δυνατότητε των ε, παρόχων υπηρεσιών ίντερνετ και να εφαρμοστούν καλύτερα τα πνευματικά δικαιώματα καταπολεμώντας ε, τις παραβιάσεις μεγάλων διαστάσεων. Έχω διάφορες ιδέες για τις τροπολογίες, αλλά όπως ξέρετε οι γνωμοδοτήσεις πρέπει να έχουν περιορισμένο μήκος. Προβλέπω να προτείνω τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης όσον αφορά τις διακρίσεις, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ τιμών, να ενισχύσουμε την ενίσχυση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρετε ποιες είναι οι ουσιώδεις προτεραιότητες. Η δημιουργία ενός καλύτερου νόμικου πλαισίου για τη δραστηριότητα στον τομέα αυτό, τον ψηφιακό και πιο συγκεκριμένα το θέμα της προστασίας των διανοητικών δικαιωμάτων. Η αγορά αυτή έχει τζίρο 450 δισεκατομμύρια ετησίως και θα μπορούσε να δημιουργήσει πολύ καλύτερες ψηφιακές υπηρεσίες. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για τα θέματα αυτά, καινοτόμε προσεγγίσεις και θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη να ενημερωθούν οι κανόνες για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν θέλουμε μία ανεπτυγμένη ψηφιακή αγορά και καινοτόμο πρέπει να είναι συμβατά τα συστήματά μας ούτως ώστε αυτή η αγορά να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της. Και τέλος θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι θα τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα διότι αναμένουμε την οριστική απόφαση της Επιτροπής να δούμε δηλαδή εάν ε, η Επιτροπή μας θα έχει συναρμοδιότητα για το θέμα αυτό. Προσβλέπω λοιπόν στα σχόλιά σας και πιστεύω ότι θα είναι πολύ επικοδομητικός ο διάλογος αύριο με τους ε, σκιώδες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you as well, Mr. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Ράβιεφ. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι η οικονομία που θα δημιουργηθεί από την ψηφιακή οικονομία και από τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής είναι πολύ σημαντική πηγή εσόδων. Γνωρίζουμε ότι η επιτυχία αυτής της ενιαίας αγοράς μπορεί να συνεισφέρει δισεκατομμύρια ευρώ ετησίων και να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει διαφορετική νομοθεσία όσον αφορά τα συμβατικά δικαιώματα, την ε, μεταφορά περιεχομένου, τα διάφορα επίπεδα ε, διαμεθοριακών ε, μεταφορών, καθώς επίσης και κάποιες διαφορές όσον αφορά τις τιμές και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, τα οποία διέπουν την αγορά, καθώς και διαφορετικούς κανόνες για το ΦΠΑ διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες και δεν μπορούμε να προλάβουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης αυτής της αγοράς. Θεωρούμε λοιπόν ότι η στρατηγική θα πρέπει να καθορίζει πολύ συγκεκριμένε και στοχευμένες δραστηριότητες προς τη σωστή κατεύθυνση. Η προστασία των χρηστών και κάποια ενερμονισμένα δικαιώματα θα συνεισφέρουν τη μεγαλύτερη ασφάλεια των χρηστών, κυρίως για τα διαδικτυακά συμβόλαια και το ε, διαμεθοριακό εμπόριο. Ελπίζουμε ότι τα εθνικά καθεστώτα ε, στον τομέα αυτό θα μειωθούν οι διαφορές και θα ληφθούν και κάποια περαιτέρω μέτρα προκειμένου να ενερμανίσουμε το ευρωπαϊκό δίκαιο όσον αφορά τις πωλήσει. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουν καλύτερη πρόσβαση στο πολιτιστικό περιεχόμενο ε, διαδικτυακά, γεγονός το οποίο θα επιτρέψει να υπάρχει και πολιτιστική ποικιλομορφέα στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Η κυρία Ρέντα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως αναφέραν ήδη οι συνάδελφοι, υπάρχουν κάποιες πάρα πολύ σημαντικές επιτυχίες της στρατηγικής ε, για την ε, εσωτερική ψηφιακή αγορά. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω κάποιες από αυτές ο στόχος ε, της ψηφιοποίησης της ε, ψηφιακής αγοράς ε, δεν μπορεί να γίνει χωρίς να λάβουμε υπόψη κάποια ζητήματα που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και για την ομάδα μου σημαντικό είναι να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί η διασυνοριακή πρόσβαση στα πολιτισμικά αγαθά στον εμπορικό αλλά και μη εμπορικό χώρο, για παράδειγμα δημόσια, δημόσια μετάδοση. Επίσης, ο κανονισμός για τα ψηφιακά μέσα που έχουμε πρέπει να συμπεριλάβει και τα δικαιώματα του κοινού. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια της στρατηγικής για την ψηφιακή εσωτερική αγορά κάτι το οποίο έχουμε εντοπίσει και σε αρκετές εκθέσεις σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και κάτι που συζητούμε σε αυτήν την Επιτροπή τελευταία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο όταν όταν πολλές φορές ασχολούνται με περιπτώσεις όπου ζητείται περισσότερη ανάληψη ευθυνών και ταυτόχρονα περισσότερη ανεξαρτησία και ουδετερότητα. Όταν ζητά σε κάποιον να είναι ουδέτερο, του ζητά ταυτόχρονα να λαμβάνει και ε, αποφάσει οι οποίε ε, είναι πιο απομακρυσμένες από τις πραγματικές ανάγκες. Όταν όμως τους ε, ζητάς να αναλάβει περισσότερες ευθύνες, τους ζητάς να είναι και περισσότερο υποκειμενικός. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μία εκ νέου αξιολόγηση της ψηφιακής μας στρατηγικής. Ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν η τελευταία που ζήτησε το λόγο. Μπορούμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό της ημερησίας διάταξης, εκτός και αν ο κύριος Τζάμπασης θέλει να προσθέσει κάτι. Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με το σημείο 32. για την εξέταση του σχεδίου εξουσιοδότηση της Αυστρίας, Βελγίου και Πολωνίας να κυρώσουν τη σύμβαση της Βουδαπέστης για τις συμβάσεις εμπορευματικών μεταφορών μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών ή να προσχωρήσουν σε αυτή. Η είμαι εγώ, μου δίνω λοιπόν το λόγο και προτείνω το Κοινοβούλιο να δώσει τη συγκατάθεσή του στην προσχώρηση σε αυτήν την σύμβαση για τις χώρες αυτές. Η σύμβαση αυτή συνεισφέρει στην εσωτερική αγορά, στον τομέα των ε, ε, μεταφορών εναρμονίζοντας τα πρότυπα για τις εμπορευματικές μεταφορές μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών. Το άρθρο 29 περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την επιλογή νομοθεσίας από τα συμβαλόμενα μέρη της σύμβασης και αυτές οι διατάξεις επηρεάζουν επομένως τους κανόνες τους, οι οποίοι επιβλήθηκαν από τον κανονισμό Ρώμη 1. Η σύμβαση της Βουδαπέστης λοιπόν, αφορά αποκλειστικές αρμοδιότητες ε, που θα έχει η Επιτροπή. Όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο δεν μπορεί να προσχωρήσει σε αυτή τη σύμβαση. Τα κράτη-μέλη όμως μεμονωμένα μπορούν, έχοντας προηγουμένως λάβει την ε, έγκριση. Ε, Και στην περίπτωση αυτή η αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζεται σε μία μόνο διάταξη, την εξουσιοδότηση δηλαδή στα ε, κράτη-μέλη και δεν θα έχει κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στην εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης για τη δικαστική συνεργασία σε αστικά και εμπορικά ζητήματα. το σχέδιο απόφαση λοιπόν εξουσιοδοτεί την Αυστρία και το Βέλγιο, την ε, το Βέλγιο και την Πολωνία να ε, προσχωρήσει και την Αυστρία να αποχωρήσει από αυτήν τη σύμβαση. προθεσμία είναι... Το μεσημέρι λοιπόν και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος από εσάς θέλει να λάβει το λόγο. Δεν βλέπω να υπάρχει κανείς. Και συνεχίζω λοιπόν με το σημείο 33. Ωστόσο, μας λείπει η συγγήτρια, η κυρία Φεράρα. Α, μόλις προλάβατε. Καλώς ήρθατε. We are just at point number... Είμαστε στο σημείο 33. Μία πρόταση δική σας για οδηγία του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2011 κάθετος 16 σχετικά με την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον χώρο της φορολόγησης. Και έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά πολλές φορές ε, υπάρχουν αλληλοκοπαλήψει μεταξύ των επιτροπών και είναι δύσκολο να είμαστε ταυτόχρονα σε όλα τα σημεία. Το Σουηδικό Κοινοβούλιο έστειλε μια αιτιολογημένη γνώμη για την πρόταση οδηγία, ε, για την τροποποίηση τη οδηγία του 2011-16 για την αυτόματη ανταλλαγή ε, πληροφοριών και ω αρμόδια επιτροπή και βάσει τις αρχές της επικορικότητας πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα αυτό, αλλά δυστυχώς η γνωμοδότηση που έλαβα είναι στα Σουηδικά. Πρόκειται για μια γλώσσα την οποία δεν κατέχω, επομένως δεν κατάφερα να λάβω ε, καν ε, μετάφραση. Ε, συγγνώμη. Ζητούν να μιλάτε λίγο πιο αργά. Ναι, εντάξει, θα τα πω πιο αργά. από τη γραμματεία μου λένε ότι το θέμα το οποίο φύγει το Σουηδικό Κοινοβούλιο είναι ότι η πρόταση οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπερβαίνει τα απαραίτητα όρια για την ε, υλοποίηση του στόχου. Ε, Ιδίω όταν ζητά από τις αρχές των κρατών μελών να παρέχουν φορολογικές πληροφορίες μέχρι και 10 χρόνια πριν. Ε, βεβαίως πριν προχωρήσει η διαδικασία της αρμοδιότητές μας επιφυλάσσομαι ώστε να λάβω και το κείμενο του Συνδικού Κοινοβουλίου μεταφρασμένο στα Ιταλικά για να μπορέσω να εκφράσω και την άποψή μου. Επί της ουσίας. Ευχαριστώ πολύ. So, uh, Επομένως αναβάλουμε το σημείο αυτό για μια άλλη συνεδρίαση. Ωραία. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την ημερήσια διάταξη. Να σας πω απλώς ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων θα γίνει στις Βρυξέλλες στις 13 Ιουλίου και 14 Ιουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας σήμερα. Είστε επανειδή.